Ladies and gentlemen. Σας ευχαριστώ πολύ κυρίες και κύριοι. Ως νέα πρόεδρος της Επιτροπής ε, ΡΕτζη, Είμαι, είναι μεγάλη τιμή μου που σας καλωσορίζω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και που χαιρετώ τον Πρόεδρο της Επιτροπής των Περιφερειών, κύριο Μισελ Λεμπρά, και τον Επίτροπα για την Περιφερειακή Πολιτική, Γιωχάνες Χάν. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Χάν για την συνεχή του δέσμευση και συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ακόμα και τον Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαφωνούσαν στο παρελθόν. Αυτός φάνηκε πολύ ισχυρός και ανοιχτός εταίρος. Ελπίζουμε ειλικρινά να παραμείνει υπέρμαχος της πολιτικής συνοχής και στους μελλοντικούς του ρόλο, στα μελλοντικά του καθήκοντα. Το αποτέλεσμα των ευρωπαϊκών εκλογών το Μάιο είχε ως συνέπειο ότι η σύνθεση της Επιτροπής μας άλλαξε δραματικά. Είμαι όμως βέβαιη ότι κι εσείς ε, θα καλωσορίσετε όπως κι εγώ την επιστροφή κάποιων από των πλέον έμπειρων μελών μας και θα τους ευχηθείτε κάθε επιτυχία στις, στα, και θα ευχηθείτε κάθε επιτυχία στους νέους συναδέλφους. Τα νέα μέλη συμπεριλαμβάνουν και δύο πρώην μέλη της Επιτροπής των Περιφερειών, την κυρία Μπρέσο και τον κύριο Βαλικαρσέλη. Άσχετα όμως αν έχουμε ήδη εμπειρία ως ευρωβουλευτές, αν είμαστε πρώην μέλη της Επιτροπής των Περιφερειών ή εντελώς καινούργιες στις Βρυξέλλες, έχουμε ένα πράγμα κοινό. Όλοι θέλουμε να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη της πολιτικής συνοχής. Σε έναν καιρό οικονομικής δυσκολίας, η πολιτική συνοχής παίζει κρίσιμο ρόλο προκειμένου να δοθεί νέο και νέα κινήτρα στην οικονομική μηχανή της Ευρωπής. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε φιλόδοξοι και θα πρέπει να υπάρξουν αποτελέσματα από την πολιτική συνοχή. Και θα πρέπει η χρήση των βέλτιστων πρακτικών να καθοδηγεί την εφαρμογή της. Σήμερα έχουμε την ε, χαρά να καλωσορίσουμε τον πρόεδρο του ΑΣΕ, Άγγελ Κουρία, ο οποίος θα μας ε, πει πώς οι άλλες περιφέρειες του κόσμου ε, θεωρούν την ε, Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνοχής και πώς εμπνέονται από αυτή. Κυρίες και κύριοι, μπορούμε να είμαστε περήφανοι από τα αποτελέσματα που έχουμε πετύχει ως τώρα. Αλλά δεν μπορούμε να αρκεστούμε απλά στις ε, επιτυχίες του παρελθόντος. Ιδιαίτερως η Επιτροπή Ρέτζη θα χρησιμοποιήσει το κοινοβουλευτικό της δικαίωμα για να ζητήσει πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να διασφαλίσει ότι η εφαρμογή της νέας ε, νομοθεσίας για την συνοχή θα περάσει από προσεκτικό έλεγχο. Οι πιο συχνέ ε, αναφορέ στην Επιτροπή Ρέτζη ήταν ένα από τα βασικά ζητήματα τα οποία έθεξαν τα μέλη μα σε πρόσφατη ακρόαση του υποψηφίου της υποψηφία ε, Επιτρόπου για την Περιφερειακή Πολιτική τη Κυρία Κρέτου. Και αυτό δεν πρόκειται να το ξεχάσουμε. Η Επιτροπή λοιπόν θα πρέπει να περιμένει ότι η Επιτροπή Ρέτζη θα επιμείνει σε ό,τι αφορά θέματα έγκαιρης και αποτελεσματικής εφαρμογής. Θα επισκεφτούμε τα κρατημέλη για να ελέγξουμε και να παρακολουθήσουμε την εφαρμογή επιτόπου. Θα ε, θέσουμε ερωτήματα στην Επιτροπή αν η πρόοδος καθυστερήσει και θα διοργανώσουμε ακροάσεις για να ενημερώσουμε τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τους εμπλεκομένους φορείς γιατί οι πολίτες μας θέλουν αποτελέσματα να δουν. Θα πρέπει να συνεργαστούμε με ξεχωριστούς αλλά συμπληρωματικούς ρόλους για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα τους απογοητεύσουμε. Δεν θα απογοητεύσουμε τους πολίτες της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Λεμπρά, τον πρόεδρο της Επιτροπής των Περιφερειών. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Επίτροπε, κύριε Γενική Γραμματέα του ΟΣΑ, κυρίες και κύριοι, εκφράζω την χαρά μου για την έναρξη των εργασιών αυτών γίνεται για μια ακόμη φορά στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που το ευχαριστώ που μας υποδέχθηκε. Η συνάντησή με σήμερα δεν είναι η συνέχιση απλά μιας παράδοσης. Είναι κάτι το οποίο συμπίπτει και με το τέλος της διαδικασίας των ακροάσεων για τους υποψηφίους επιτρόπους, με μια νέα κοινοβουλευτική περίοδο και με ένα νέο θεσμικό πλαίσιο. Θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω, να σας ευχαριστήσω αγαπητέ Ραμόν Λουίς και κυρία Μιχαήλοβα γιατί για μια ακόμη φορά οργανώσατε την κοινή συνάντηση των Επιτροπών Ρίτζι και Κότερ των δύο οργάνων, του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής των Περιφερειών. Ο Επίτροπος ο υπεύθυνος για τα θέματα της περιφερειακής πολιτικής ε, όχι μόνο σημαδέψατε την πολιτική μας κύριε Χάν, αλλά σημαδέψατε και αυτήν την συνάντηση η οποία για δωδέκατη φορά οργανώνεται. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών υπήρξαν πολύ σημαντικές αλλαγές στα πλαίσια της διακυβέρνησης της ευρωπαϊκής πολιτικής και της περιφερειακής πολιτικής. Υπό την αιγίδα σας κύριε, Χάν έγινε η περιφερειακή πολιτική μια πολιτική επενδυτική συνδεδεμένη άμεσα με αποτελέσματα και επίσης άμεσα συνδεδεμένη με τη νέα οικονομική διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με την Ευρώπη του 2020. Έχει φτάσει η στιγμή των συγκεκριμένων πλέον επιτευγμάτων και αυτός θα είναι και ο καρπός των συνεδριάσεών μας σήμερα. Θα πρέπει να προσφέρουμε στη χρηματοδότηση των πόλεων μας, των περιφερειών μας, να προχωρήσουμε σε ευφυείς μορφές επένδυσης προς το συμφέρον των πολιτών. Αυτό είναι το πρόγραμμα δράσης των νέων προγραμμάτων στα πλαίσια της νέας προγραμματικής περίοδου 2014-2020. Εξ ονόματος όλων των συμμετεχόντων σας ευχαριστώ κύριε Χάν, κύριε Επίτροπε για όλα αυτά τα χρόνια που σταθήκατε αρρωγός στις περιφέρειες και που σταθήκατε εκεί για να μας βοηθήσετε και να καλύψετε τις ανησυχίες μας. Κύριε Γκουρία, Γενική Γραμματέα του ΟΣΑ, θα ήθελα να, ευχαριστήσω, να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Νομίζω ότι δεν κάνω λάθος όταν λέγω ότι η Επιτροπή Περιφερειών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμερίζονται την ίδια ανάλυση του ρόλου των ευφυών δημοσίων επενδύσεων που είναι απαραίτητες για να καλύψουν τις ανάγκες που έχουν οι οικονομίες μας και οι αγορές εργασίας μας στον δρόμο της ανάπτυξης και της βελτίωσης της ανθεκτικότητάς τους. Σας ευχαριστώ επίσης που στα πλαίσια αυτών των Open Days θα μας παρουσιάσετε και τα πρώτα συμπεράσματα των περιφερειακών πολιτικών 2014 του ΟΣΑ, όπως επίσης και την έκθεση για την λεγόμενη ευημερία των περιφερειών. Κύριε Γκουρία, να σας ευχαριστήσω και για το μνημόνιο συνεργασίας που υπογράψαμε εσείς για τον ΟΣΑ και εγώ για την Επιτροπή των Περιφερειών για να ενισχύσουμε την συνεργασία μας η οποία ήταν ήδη αποτελεσματική. Κυρίες και κύριοι, με την ευκαιρία αυτή να αναφέρω ότι το πρόγραμμα αυτών των ημερών προέρχεται από την συνεργασία 200 πόλεων και περιοχών από 30 χώρες, από τη συνεργασία 11 Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πολλαπλών δικτύων και ενώσεων ευρωπαϊκών. Πολλοί από όλου αυτούς είναι παρόντες σήμερα, όχι όμως όλοι. Τους ευχαριστώ όλους για την υποστήριξή τους. Θα ήθελα επίσης ε, ένα τελευταίο λόγο να πω προς τους ε, άμεσα στους ερετούς ε, της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Συνάδελφοι, η Επιτροπή των Περιφερειών είναι το δικό σας όργανο. Έχει σαν στόχο να ε, συμβουλεύει τα ευρωπαϊκά όργανα γύρω από θέματα περιφερειακής και τοπικής πολιτικής. Εμείς προσπαθούμε λοιπόν να μεταφέρουμε τις απόψεις σας στο επίπεδο το ευρωπαϊκό. Προσπαθούμε να προασπιστούμε την διακυβέρνηση, την πολυεπίπεδη και την επικουρικότητα στα πλαίσια της ε, περιφερειακής πολιτικής. Ο ρόλος αυτός είναι απαραίτητος γιατί η Ευρώπη αλλάζει. Η Ευρώπη ξεκινά μια νέα νομοθετική περίοδο και αυτές οι αλλαγές θα τροφοδοτήσουν τις συζητήσεις τους επόμενους μήνες. Να είστε σίγουροι ότι θα αναλύσουμε τις προτάσεις σας αυτές σε βάθος και η φωνή σας, η δική μας φωνή, θα ακουστεί έτσι ώστε να ληφθούν υπόψη οι ανησυχίες σας σας καλώ να είστε σε μόνιμη επαφή με την Επιτροπή των Περιφερειών, όχι μόνο κατά τη διάρκεια αυτών των συναντήσεων. Κλείνοντας, να σας ευχηθώ λοιπόν, καλώς ορίσατε και δίνω αμέσως το λόγο στον πρώτο μιλητή μας, τον Ραμόν Λουίς Βαλκάρσελ Σίσο. Είσαστε, θα έλεγα, στην καλύτερη θέση σαν τελευταίος πρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών και νυν αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να αναγνωρίσετε τον ρόλο και τη σημασία των πόλεων και των περιφερειών ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε λοιπόν την άποψή σας και σαν νέου Ευρωβουλευτή, ε, άλλωστε εσείς εκπροσωπείτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σήμερα. Σας ευχαριστώ. Και τώρα έχω την τιμή να δώσω το λόγο για την βασική ομιλία στον Ραμόν, στον κύριο Ραμόν Λουίς Βαλκαρσέλ Σίσο, αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχετε το λόγο. Πρόεδρε της Επιτροπής ε, Περιφερειακών Υποθέσεων, κυρία Μιχαήλοβιτς, αγαπητέ Μισελ Λεμπρά, αγαπητέ κύριε Γκουρία, αγαπητέ κύριε Επίτροπε Χάν, αγαπητοί συνάδελφοι, φίλοι, σας φαίνονται λίγο τυπικά όλα αυτά, αλλά θα ήθελα να πω ότι το κάνω όλο εγκαρδίως, γιατί είναι τιμή μου που είμαι σήμερα στην έναρξη μιας συνεδρίασης όπως αυτή, τα Open Days δηλαδή, γιατί μου δίνουν την ευκαιρία να συναντηθώ με τόσους πολλούς φίλους. Ήμουν μέλος της Επιτροπής Περιφερειακών Υποθέσεων ε, για πάνω από 20 χρόνια και μέχρι πριν λίγους μήνες πρόεδρος της οργάνωσης αυτής και συνειδητοποιώ την προσπάθεια η οποία γίνεται εδώ για να καλυφθούν τα συμφέροντα των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι θα έλεγα μια εξαιρετική ε, ευκαιρία να ανταλλάξουμε εμπειρίες και να δούμε τις επιπτώσεις της πολιτικής, της περιφερειακής και της πολιτικής συνοχής και είναι μια κατάλληλη στιγμή για να ενισχύσουμε το, τα ευρωπαϊκά προγράμματα και να καλύψουμε τις προσδοκίες του Ευρωπαίου πολίτη. Η συνεργασία ανάμεσα στα θεσμικά όργανά μας ήταν πάντα το κάτι πολύ σημαντικό και η συμφωνία που υπεγράφει τον μήνα Φεβρουάριο δεν είναι παρά η κορύφωση αυτής της συνεργασίας. Δείχνει τη μεγάλη σημασία που δίδουμε στην επικουρικότητα και στην λεγόμενη πολυεπίπεδη διακυβέρνηση στα πλαίσια ο καθένας των αρμοδιοτήτων του. Έτσι λοιπόν αυτός ο διοργανικός διάλογος αντικατοπτρίζει τα συμφέροντα και τις προσπάθειες και των δύο οργάνων για να προωθήσουν τις αρχές ε, του βασικού πυλώνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι η περιφερειακή πολιτική. Ο συνδυασμός των, ε, δύο οργάνων της Επιτροπής των Περιφερειών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ενισχυθεί αυτό φαίνεται και από τις εκθέσεις μας και από τους εισηγητές που έχουμε επιλέξει. Και νομίζω ότι έτσι θα επηρεάσουμε με σωστότερο τρόπο την τελική διατύπωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή των Περιφερειών θα κάνουμε κάθε προσπάθεια έτσι ώστε να ληφθούν οι επιθυμίες σας υπόψη. Κυρίες και κύριοι, κύριε Χάν, αγαπητέ Γιωχάνες, θα ήθελα για μια ακόμη φορά να αναγνωρίσω την τεράστια προσπάθεια που έκανε σαν επίτροπο στο επίπεδο της περιφερειακής πολιτικής όλα τα τελευταία χρόνια. Ήσασταν πάντα ένας υπερασπιστής της περιφέρειας σε όλα τα όργανα τα ευρωπαϊκά και σε όλα τα επίπεδα και χρησιμοποιήσαμε και μείναμε στην πολιτική αυτή όταν πολλοί είχαν αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα της πολιτικής αυτής ιδιαίτερα μετά από τις μακροοικονομικές συνέπειες που είχαν προκληθεί λόγω της κρίσης. Η Ευρώπη θα πρέπει εκ νέου να στέλνει σήματα οικονομικής ανάκαμψης. Η ανάκαμψη αυτή όμως δυστυχώς δεν έχει εμποδίσει οι διαπεριφερειακές ανισότητες να αυξάνονται, όπως το δείχνει άλλωστε και η έκθεση για την οικονομική και εδαφική συνοχή. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν θα πρέπει να ενισχύσουμε την περιφερειακή διάσταση των ευρωπαϊκών πολιτικών. Έχει μεγάλη σημασία όλοι να εργαστούμε για να δώσουμε εγγυήσεις για μια σωστή πολιτική συνοχής, αντίστοιχη με τις ανάγκες των περιφερειών μας γιατί η περιφερειακή πολιτική είναι το καλύτερο μέσο που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να καλύψει τον δρόμο που θα οδηγήσει στην οικονομική ανάκαμψη και στη δημιουργία απασχόλησης. Μια πραγματική περιφερειακή πολιτική θα πρέπει να εφαρμοστεί και στον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στην καινοτομία και στην ενέργεια Αυτά τα πλαίσια αποτελούν μια πηγή δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, όπως οι πράσινες θέσεις απασχόλησης, η κάλυψη της ζήτησης ειδικευμένου προσωπικού στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας των τηλεπικοινωνιών και την ενίσχυση ενός προτύπου ανάπτυξης αηφόρου και χωρίς αποκλεισμούς. Αυτός είναι όπως είχε πει και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο νέος ε, ο στόχος του ο βασικός, δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Αυτός είναι ο κοινός στόχος που πρέπει όλοι να επιδιώξουμε. Πρέπει ο Ευρωπαίος να νιώθει την Ευρώπη δίπλα του. Είναι επίσης απαραίτητο να θέσουμε σε λειτουργία ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανάπτυξης που να δίνει κίνητρα στην επενδύσεων, πρόγραμμα που να δίνει κίνητρα στην πολιτική ανάκαμψη. Γιατί καμιά φορά ανησυχώ, γιατί στην Ευρωπαϊκή Ένωση μερικές φορές βάζουμε και κάποια εμπόδια στην ανάκαμψη των περιφερειών και αυτό για πολλούς λόγους. Πρέπει σίγουρα να εφαρμόσουμε την μέγιστη δυνατή υπαρκτή σήμερα ευελιξία για την σωστή χρήση των περιφερειακών ταμείων χωρίς καθυστερήσεις. Και αυτό θα το επιδιώξει και το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή Περιφερειών. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται πάντα με το θέμα της δημόσιας, της εθνικής συγχρηματοδότησης. Η Ιταλική Προεδρία άλλωστε του Συμβουλίου έχει θέσει το θέμα αυτό και το έχει καταστήσει μια βασική της προτεραιότητα. Ελπίζουμε να υπάρξει μία σύντομα μία απάντηση σε αυτό. Οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές ξέρουν ότι μπορούν να θεωρούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σαν σύμμαχό τους και για το θέμα αυτό. Δεύτερον, μας ανησυχεί και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι καθυστερήσεις πληρωμών που συνδέονται με την πολιτική συνοχής. Στο τέλος του προηγούμενου χρόνου τα μη πληρωμένα αλλά ε, οι, πιο, ε, οι μη πληρωμένες δαπάνες έφταναν ε, πάνω από 13 δις. Νομίζω ότι αυτά όλα δημιουργούν πάρα πολλά προβλήματα ιδιαίτερα στις περιοχές οι οποίες θίγονται από την οικονομική κρίση. Θα πρέπει να μειώσουμε τις καθυστερήσεις και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δώσουμε λύσεις στα προβλήματα αυτά ε, το ταχύτερο δυνατόν σε συνεργασία με την Επιτροπή. Θα ήθελα επίσης κυρίες και κύριοι οι περιφέρειες να καθορίσουν σωστά τις σχέσεις του με τις πρωτεύουσες των χωρών στις οποίες βρίσκονται για να μην υπάρχουν περαιτέρω καθυστερήσεις. Θεωρώ ότι για να εκμεταλλευτούμε σωστά τον πλούτο των περιφερειών μας όχι μόνο θα πρέπει να χρησιμοποιούμε δείκτες που εξχετίζονται με το ΑΕΠ της κάθε χώρας, αλλά και άλλους δείκτες που αντικατοπτρίζουν ίσως καλύτερα τις ανάγκες και την ποιότητα της ζωής των πολιτών. Και γι' αυτό εδώ αναγνωρίζω την εξαιρετική εργασία που έχει κάνει ο ΩΣΑ, του οποίου ο Γενικός Γραμματέας σήμερα μας κάνει την τιμή να είναι παρόν και θα μας δώσει την δυνατότητα να γνωρίσουμε καλύτερα την πραγματικότητα των περιφερειών μας. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο για τις εργασίες σας. Thank you, Mr. Σας ευχαριστώ κύριε Βαλκαρσέλ και τώρα δίνω το λόγο στον Επίτροπο για την Περιφερειακή Πολιτική, στον Γιωχάννη Χάν. Έχετε το λόγο. <clears throat> Um, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρόεδρε, ε, Αντιπρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, φίλοι της περιφερειακής πολιτικής. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω όλους σήμερα Να σας καλωσορίσω ιδιαίτερα φέτος ε, στα Open Days, διότι για μένα είναι ιδιαίτερα σημαντική στιγμή. Άλλωστε είναι η τελευταία φορά που συμμετέχω ως επίτροπος αρμόδιος για την περιφερειακή πολιτική στα Open Days. Θυμάμαι πολύ καλά την πρώτη φορά το 2010. Τότε αρχίσαμε να νιώθουμε τις ε, επιπτώσεις ε, της κρίσης ε, και μόλις είχε δημοσιευτεί η πέμπτη έκθεση συνοχής και ήταν η έναρξη της περίοδου προβληματισμού για την πολιτική συνοχής. Ήδη ήταν σαφές ότι η περιφερειακή πολιτική δεν μπορούσε να συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο. Και θυμάμαι ότι στην ομιλία μου ανέφερα τρεις σημαντικές πτυχές της μελλοντικής πολιτικής συνοχής. Συγκέντρωση, αποτελέσματα και προϋποθέσεις το 2010 υπήρχε αρκετό σκεπτικισμός σχετικά με την προστιθέμενη αξία της πολιτικής συνοχής και η καλύτερη απάντηση στις επικρίσεις ήταν μια μεταρρύθμιση της πολιτικής συνοχής ώστε να γίνει ένα πραγματικό εργαλείο στρατηγικών επενδύσεων για τις περιφέρειες ώστε να πετύχουμε τους στόχους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα που πλησιάζει το τέλος της θητείας μου Ω Επίτροπος ε, της περιφερειακή Πολιτικής ε, δεν θέλω να κρύψω την υπερηφάνειά μου. Νιώθω σαν ένας πατέρας που βλέπει το παιδί του να μεγαλώνει. Διότι πέντε χρόνια μετά έχουμε πράγματι μια μεταρρυθμισμένη πολιτική συνοχή που είναι πιο στρατηγική, πιο επικεντρωμένη και πιο προσανατολισμένη στα αποτελέσματα. Παρέχει το ε, σωστό πλαίσιο για αποτελεσματικέ επενδύσει στις περιφέρειές μα και συμβάλλει στον στους στόχους ε, της Στρατηγικής Ευρωπαϊκή Ένωση 2020. Ω αποτέλεσμα της μεταρρύθμισης έχει αλλάξει και η νοοτροπία των ανθρώπων. Η πολιτική συνοχής δεν θεωρείται πια ένα, ένα ταμείο από χρήματα που ε, απλά πρέπει να μοιραστούν. Ε, η φιλοσοφία των επενδύσεων γίνεται περισσότερο αντιληπτή και αυτό δεν οφείλεται μόνο στην αλλαγή της ονομασίας των Ευρωπαϊκών και Επενδυτικών Ταμείων, αλλά οφείλεται στην μεταρρύθμιση που δίνει προτεραιότητα στην στρατηγική ε, και όχι στα ε, μεμονωμένα προγράμματα. Βρισκόμαστε τώρα στην αρχή τη ε, περίοδου 2014-2020. Είναι το πιο κρίσιμο στάδιο, διότι αυτή τη στιγμή καθορίζουμε το πλαίσιο για την δαπάνη των ταμείων. Οι διαπραγματεύσεις θα οδηγήσουν σε ολοκλήρωση των σχετικών εγγράφων και η Κομισιόν μέχρι σήμερα έχει οθετήσει 16 Πιθανότατα ε, άλλη μια συμφωνία ε, αυτή την εβδομάδα με τη Φιλανδία. Ε, στο τέλος εβδομάδας θα έχουμε συνάψει 17 συμφωνίες εταιρικής σχέσης που αντιπροσωπεύουν επάνω από 300 δισεκατομμύρια ευρώ ε, που αντιπροσωπεύουν το 70% του ε, συνολικού προϋπολογισμού των ε, διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων. Έχουμε λάβει το 95% των προγραμμάτων, αλλά μέχρι στιγμής έχουμε υιοθετήσει μόνο, δύο, μόνο 7. Απομένουν πολλά να γίνουν ακόμα. Θα πρέπει να επενδύσουμε σε προγράμματα και στην πραγματική οικονομία. Ωστόσο, δεν θα πρέπει η ποιότητα μάλλον η ταχύτητα να είναι εις βάρος της ποιότητας. Άλλωστε, αυτά αποτελούν τον προγραμματισμό για την επόμενη επταετία και αν λάβουμε υπόψη τις προϋποθέσεις, μιλάμε για την επόμενη δεκαετία. Με την πρώτη ανάλυση των πληροφοριών έχουμε λάβει πολύ ενθαρρυντικά ε, μηνύματα σχετικά με το πώς θα μεταφέρουμε την ε, μεταρρύθμιση στην πράξη. Για παράδειγμα, είναι ήδη σαφές ότι τουλάχιστον 125 δις θα κατανεμηθούν για να υποστηριχθούν οι επιχειρήσεις, η έρευνα και ανάπτυξη, η καινοτομία, οι τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών, καθώς και η οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξείδιου του άνθρακα. Αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση πάνω από 20% σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα, κάτι που αντικατοπτρίζεται με ανάλογη μείωση στην ε, υποστήριξη για τις υποδομές. Φυσικά θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την ανάπτυξη υποδομών στα περισσότερα κράτη-μέλη. Η διαφορά αυτή τη φορά είναι ότι κάνουμε πιο στρατηγική επιλογή των προγραμμάτων που θα συμβάλλουν σε έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη. Θέλουμε να δημιουργήσουμε βιώσιμες δυνατότητες για τις επιχειρήσεις και αυτό και θέσεις απασχόλησης. Ε, έτσι θα αντιμετωπίσουμε το θέμα της διαρροής εγκεφάλων. Ο κόσμος θα σταματήσει να φεύγει εάν έχει ευκαιρίες στον τόπο διαμονή του και έτσι ε, το brain drain θα γίνει brain circulation, κυκλοφορία εγκεφάλων. Άλλο ενθαρρυντικό ε, σημάδι είναι ότι τα χρηματοδοτικά μέσα έχουν τώρα μεγαλύτερη σημασία. Είδαμε αύξηση στο δεκαπλάσιο από το 2000-2006 ε, μέχρι το διάστημα 2007-2013. 12,6 δισεκατομμύρια ευρώ είχαν ε, δοθεί ε, μέχρι το τέλος του 2012 σε 25 κράτη-μέλη. Στην προηγούμενη περίοδο το αντίστοιχο ποσό ήταν 1 δις ευρώ. Αναμένεται ότι για το διάστημα 2014-2020 θα δούμε υπερδιπλασιασμό της, του ποσού αυτού και θα, θα φτάσουμε τα 30 ή ακόμα καλύτερα 40 δισεκατομμύρια ευρώ. Κατόπιν έχουμε τα συγκεκριμένα μέτρα για την πρόθεση της απασχόλησης, ε, την βελτίωση των δεξιοτήτων των ανθρώπων και τη μείωση της φτώχειας. Οι αναλύσεις μας δείχνουν ε, ότι σχεδόν 100 δισεκατομμύρια ευρώ θα επενδυθούν στους ίδιους τους ανθρώπους ε, μέσα στο νέο διάστημα. Αυτό θα γίνει με μια προσέγγιση με την οποία αντιστοιχίζονται καλύτερα οι δεξιότητες με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Και έτσι θα συνδυάσουμε διάφορες πολιτικές, ε, ταμεία και προτεραιότητες. 88 προγράμματα σε 16 χώρες θα ε, χρηματοδοτηθούν από διάφορα ταμεία. Ιδιαίτερα με ενθαρρύνουν ε, οι πιστώσεις για την η οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Είναι ένας από τους τέσσερις τομείς ε, θεματικής ε, συγκέντρωσης ε, και με βάση με αυτήν τη βάση οι ελάχιστε πιστώσει θα ανέρχονταν σε 23 δισεκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, με την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργεια. Έχουμε τονίσει ένα θέμα το οποίο θα είναι ακόμα πιο σημαντικό στο παρόν κλίμα και έχω να σας ανακοινώσω άλλο ένα εντυπωσιακό νούμερο. Εάν εξοικονομήσουμε το 1% της ενέργειας κάθε χρόνο στην Ευρώπη, θα μπορέσουμε να μειώσουμε τις εισαγωγές ε, φυσικού αερίου κατά 2,6% το χρόνο. Και γνωρίζετε τι σημαίνει αυτό έχοντας κατά νου την ε, παρούσα πολιτική κρίση στην Ουκρανία και αλλού. Ως αποτέλεσμα, αυτή τη, στιγμή, ε, αυτή έχουμε 38 δισεκατομμύρια ευρώ για να υποστηρίξουμε την μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα και ε, ανθεκτική στην αλλαγή του κλίματος. Ε, και αυτό γίνεται με βάση τις 16 συμφωνίες εταιρική σχέσης από τις 28. Αυτό είναι, αποτελεί σχεδόν το διπλάσιο από αυτό που είχαμε στο διάστημα 2007 με 2013. Με συγχρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα προβλέπεται ακόμα μεγαλύτερη αύξηση, αλλά μην παρασυρώμαστε. Όσο ενθαρρυντικά και αν είναι αυτά τα σημάδια, δεν αποτελούν τίποτα παραπάνω από δεσμεύσει σε χαρτί. Είναι σημαντικό να προχωρήσουμε στην εφαρμογή των προγραμμάτων και να αρχίσουμε τις επενδύσεις σε προγράμματα που θα μεταφέρουν τη θεωρία στην πράξη. Αγαπητοί φίλοι, θα ήθελα να δράξω την ευκαιρία να μοιραστώ μαζί σα του προβληματισμού μου πάνω σε κάποιε σημαντικέ προκλήσει του μέλλοντο. Όπω γνωρίζετε, η πολιτική συνοχή εξαρτάται από το οικονομικό κλίμα στο οποίο εφαρμόζεται και για τον λόγο αυτό έχουμε εισάγει έναν σύνδεσμο ανάμεσα στη νέα πολιτική συνοχή και την οικονομική διακυβέρνηση και το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Ωστόσο, δεν έχουν ρυθμιστεί ακόμα οι λεπτομέρειες και αυτή τη στιγμή επικρατεί η θέση ότι ο μόνος ρόλος της πολιτικής συνοχής Ε, είναι να αναστέλει τη χρηματοδότηση σε χώρες που δεν πληρούν τις ε, υποχρεώσεις τους. Ωστόσο αυτό είναι μόνο η μία πλευρά του νομίσματος, ε, διότι γνωρίζουμε ότι η πολιτική συνοχή μπορεί να αποτελεί και κίνητρο και κύρωση. Άλλωστε, τα ευρωπαϊκά διαφορετικά και επενδυτικά ταμεία είναι στη διάθεση των κρατών μελών για να τα βοηθήσει να πληρούν τις προϋποθέσεις τους στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου. Η πολιτική συνοχή ε, συμπληρώνει το τρίγωνο της ε, οικονομικής διακυβέρνησης ε, και η δημοσιονομική εξυγίανση και οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις θα πρέπει να ενισχύουν το ένα το άλλον. Άλλη σημαντική πρόκληση είναι η αύξηση του διοικητικού δυναμικού στις δημόσιες αρχές και σε άλλους φορείς. Το θέμα εδώ δεν είναι τόσο πολύ τα χρήματα, αλλά η δημιουργία κατάλληλων δομών και ε, των μέσων για να γίνει σωστά η δουλειά. Πρέπει να απλοποιηθούν οι κανόνες και να οικοδομήσουμε αποτελεσματικές ε, εταιρικέ σχέσεις σε όλα τα επίπεδα. Η πολιτική συνοχή παρέχει τους πόρους και τις δυνατότητες ε, για την δημιουργία μια σύγχρονη διαφανού πολιτικής δημόσιας διοίκησης. Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα κλίμα εμπιστοσύνης και υπάρχει άλλο ένα σημαντικό πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να λυθεί στο άμεσο μέλλον. Αυτό ήδη αναφέρθηκε από κάποιους από τους προηγούμενους ομιλητές. Όπως γνωρίζετε υπάρχει ένα χάσμα ανάμεσα στις ετήσιες υποχρεώσεις και τις ετήσιες πληρωμές στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώς το χάσμα αυτό ε, μεγαλώνει κάθε χρόνο και δυσκολευόμαστε ε, να τηρήσουμε τις δεσμεύσεις μας. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου η εφαρμογή προγραμμάτων στην πράξη επηρεάζεται από την έλλειψη ρευστότητας. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτήν την αναντιστοιχία ανάμεσα στις δεσμεύσεις τους και τις αποφάσεις τους σχετικά με τον προϋπολογισμό. Δεν μπορούν να περιμένουν αποτελέσματα από εμά χωρίς να παρέχουν ε, τους απαραίτητους πόρους. Καλό λοιπόν όλους σας να χρησιμοποιήσετε τις πολιτικές εξουσίες σας στα κράτη-μέλη ώστε να φροντίσετε να παρέχετε ο απαραίτητο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι προπολογισμό για τα κράτη-μέλη. Δεν είναι προπολογισμό ε, με σκοπό μόνο την κάλυψη των ε, διοικητικών δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 6% του συνολικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποιείται για να καλύψει διοικητικές δαπάνες όλων των θεσμικών οργάνων. Πάνω από το 95% του προϋπολογισμού μας επιστρέφει στα κράτη-μέλη. Ένα μικρό ποσοστό χρησιμοποιείται για δράσεις εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν λοιπόν ζητάμε χρήματα, ζητάμε επαρκή προϋπολογισμό για να μπορέσουμε να ε, τηρήσουμε τις υποχρεώσεις μας. Σας καλώ να το έχετε αυτό κατά νου και να συνεχίσετε να ασκείτε πίεση για το θέμα αυτό. Κυρίες και κύριοι, καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας μου ήμουνα υπέρ μιας ε, πιο ισχυρής ε, αστικής πολιτικής όπου είναι σημαντική η εμπλοκή των πόλεων. Χωρίς πόλεις ποτέ δεν θα πετύχουμε τους φιλόδοξους στόχους μας ε, του προγράμματος Ευρώπη 2020. Χωρίς τις πόλεις δεν θα έχουμε αποτελεσματική έξοδο από την κρίση, δεν θα έχουμε αίσθηση, αίσθημα ιδιοκτησίας ε, και οικειοποίησης ε, του ευρωπαϊκού θεματολογίου. Στο τέλος της θητείας μου ε, ως Επιτρόπου. Ε, σημειώνω ότι έχουμε ε, σημειώσει σημαντική πρόοδο. Έχουμε μια πολιτική συνοχή με ισχυρή αστική διάσταση, αλλά χρειαζόμαστε στενή συνεργασία ανάμεσα στην Ήπεθρο και τις πόλεις, διότι οι περιοχές αυτές δεν είναι ξεχωριστές η μία από την άλλη, επικαλύπτονται και ξέρουμε πώς το αντιλαμβάνεται αυτό ο κόσμος. Το γεγονός λοιπόν ότι έχουμε μια νέα αστική διάσταση αντικατοπτρίζεται στη ε, νέα περίοδο και ε, φαίνεται ότι ε, ότι το 50 με 60% του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης θα διατεθεί για τις αστικές περιοχές. 60 δισεκατομμύρια ευρώ που είναι το διπλάσιο από την ελάχιστη απέτηση του 5%. Θα πρέπει όμως να προχωρήσουμε πιο πέρα στο μέλλον. Οι δημόσιες διαβουλεύσεις, οι προοπτικές ε, μιας νέας ε, αστικής ατζέντα δείχνει ότι χρειαζόμαστε περισσότερη συμμετοχή στην ε, διαδικασία αυτή. Θα δημοσιευτεί μια λεπτομερή ε, ανάλυση της κατάστασης μέχρι το τέλος της χρονιάς και θα ήθελα να σας καλέσω να διατηρήσουμε την ε, ορμή του ε, θεματολογίου των πόλεων. Κυρίες και κύριοι, τα Open Days δείχνουν τη σημασία της κοινή διαχείρισης. Έχουν συναυτεί έτσι ισχυρές σχέσεις όχι μόνο ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη, αλλά πιο σημαντικά ανάμεσα στο εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο με τους ενδιαφερομένους. Η συμμετοχική αυτή προσέγγιση και η αρχή της ε, εταιρικής ε, σχέσης ε, αποτέλεσαν τη βάση της επιτυχίας της πολιτικής συνοχής μας. Γνωρίζω ότι τα καλύτερα μας προγράμματα και τα πιο αποτελεσματικά δίκτυα μας ε, ξεκίνησαν ε, από την εκδήλωση των Open Days. Με την αρχή της ε, μοιρασμένης διαχείρισης και την προσέγγιση της εταιρική σχέσης, η πολιτική συνοχή έχει παρουσιάσει στην πραγματικότητα αποτελέσματα. Και ακριβώς για αυτούς τους λόγους η πολιτική συνοχή μπορεί να συμβάλλει στην επίτευξη των κοινών ευρωπαϊκών μας στόχων. Κάποιοι από τους κοινούς μας στόχους, όπως είναι οι στόχοι του Ευρώπη 2020 είναι προφανείς, ε, αλλά υπάρχουν και άλλοι στόχοι. Για παράδειγμα, ε, έχουν χρησιμοποιηθεί διαρθρωτικά ταμεία για να αντιμετωπιστεί η κρίση με την υποστήριξη ε, προγραμμάτων δημοσίων επενδύσεων που αλλιώ θα είχαν καταρρεύσει και επίσης συμβάλλει στη συμπληρώση των κενών στα μεγάλα μεταφορικά δίκτυα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, και επίσης βοηθούν για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα τη ενεργειακή εξάρτηση. Η μεταρρύθμιση έχει πετύχει η πολιτική συνοχή να αποτελεί εργαλείο για να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε πρόκλησή μα από το 2020 και μετά. Αποχαιρετώντα σα, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλου του ανθρώπου που ε, ε, κατέστησαν εφικτή την μεταρρύθμιση. Ιδιαίτερα θα ήθελα να εκφράσω την εκτίμησή μου προ του συναδέλφου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή των Περιφερειών η πρώην πρόεδρος ε, της Επιτροπής Ρέτζη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η κυρία Ντανούτε Χίβνερ, ε, και ο, πρόεδρος, ε, ο πρώην πρόεδρος η πρώην πρόεδρο τη Επιτροπή των Περιφερειών ε, Μερσέντε Πρέσο και ο κύριο Ραμόν Λούι Βαλκαρσέλ έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στην μεταρρύθμιση. Θα ήθελα επίση ε, να ε, ευχαριστήσω τον Άγγελ Κοέρια για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε κατά τη διάρκεια των ετών με τον ΩΣΑ και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους ε, εσάς που αναγνωρίζω και στο κοινό σήμερα που είχα τη χαρά να συναντήσω και να συνεργαστώ μαζί τους ε, μέσα στην προηγούμενη πενταετία κατά τις επισκέψεις μου στις περιφέρειες. Εσείς είσαστε οι άνθρωποι που καταφέρατε να πετύχουν τα πράγματα επί τόπου η ανάπτυξη των ε, περιφερειών της Ευρώπης ε, είναι ένα θέμα που θα με ενδιαφέρει και στο μέλλον παρότι ε, θα αλλάξω καθήκοντα και μπορείτε να είσαστε βέβαιοι για την, τις συνεχείς προσπάθειές μου στο θέμα αυτό. Και θα ήθελα να σας καλέσω να επικεντρωθείτε στην ολοκλήρωση των, των εγγράφων προγραμματισμού. Όπως είπα πριν, μην είναι η ταχύτητα εις βάρος της ποιότητας, αλλά να αδράξετε τις ευκαιρίες που σας παρέχει η νέα πολιτική συνοχή για να κάνετε τις σωστές επενδύσεις για τις περιφέρειές σας. Θα πρέπει να μπορέσουμε να παίξουμε σημαντικό ρόλο στη ζωή των ανθρώπων. Τα τελευταία χρόνια εξαρτιόμασταν από ε, αυτούς που σχεδιάσανε την πολιτική. Τώρα όμως πρέπει να εφαρμοστεί η πολιτική αυτή. Ε, ελπίζω ε, να υποφεληθείτε από τις φετινές Open Days. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, Σας ευχαριστώ, Επίτροπε. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Ζωζέ Αγγελγκορία, Γενικό Γραμματέα του ΩΣΑ. Έχετε το λόγο. Κύριε... Αντιπρόεδρε Βαλκάσιλ, Επιτροπέ Χάν, αγαπητέ Γιωχάνες, αγαπητοί βουλευτές, κυρίες και κύριοι, συνάδελφοι και φίλοι. Χαίρομαι ιδιαίτερως που στην αρχή αυτών των ανεκτών ημερών του 2014 βρίσκω Βρίσκομαι εδώ μαζί σα, μαζί με την Επιτροπή των Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συνεργαζόμαστε εδώ και πολλά χρόνια και φυσικά θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μα για να προωθήσουμε την αποτελεσματική περιφερειακή ανάπτυξη. Πριν από κάποιες ώρες, όπως ανέφερε και ο πρόεδρος Λεμπράν, υπογράψαμε μνημόνιο συμφωνία με την Επιτροπή των Περιφερειών για να οργανώσουμε το έργο μας, αλλά και για να δεσμευθούμε στην πιο συστηματική συνεργασία στο μέλλον. Οι ανοιχτές αυτές οι μέρες λοιπόν αποτελούν μια ευκαιρία για να κοιτάξουμε τις έξυπνες επενδύσεις για τον κόσμο. Έξι χρόνια μετά την έναρξη της κρίσης ο κόσμος ζητά στην Ευρωπαϊκή Ένωση πιο πολλή ανάπτυξη, πιο πολλέ θέσει εργασία, μεγαλύτερη ποιότητα ζωή και πιο πράσινο μέλλον. Μακρύ ο κατάλογο, ίσω ε, υπερβολικά μακρύ για τις λίγες, ε, τα, τα λίγα επενδυτικά μέσα που έχουμε. Γι' αυτό λοιπόν στρατηγική επένδυση χρειάζεται αν θέλουμε πρόοδο και να πετύχουμε τους στόχους μας και να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των πολιτών. Κάποιες εθνικές κυβερνήσεις ε, είναι υπεύθυνε για το, μεγάλο, το μεγαλύτερο ποσοστό των δημοσίων επενδύσεων, για 72%. Η πίεση στις δημόσιες προπολογισμού για να διατηρηθούν οι δαπάνες σε ψηλό επίπεδο αποτελεί τη μεταβλητή προσαρμογή στα τελευταία χρόνια και ουσιαστικά μεταξύ του 2007 και το 2012 ο όγκος των υποεθνικών επενδύσεων στις χώρες ε, ε, όσα μειώθηκε κατά 4%. Θα ήθελα λοιπόν σήμερα να τονίσω κάποιες διόδους πολιτικής και κάποια εργαλεία διακυβέρνησης που χρησιμοποιούμε για να απαντήσουμε στο γιατί, πού και πώς μπορούν να είναι αποτελεσματικές μελλοντικές επενδύσεις. Και γι' αυτό λοιπόν εστιαζόμαστε στο θέμα αυτό, στις δημοσιεύσεις που παρουσιάζουμε σήμερα. Regional Outlook, περιφερειακή προοπτική για τον ΣΑΕΚ 2014 και πώς είναι η ζωή στην περιφερειά σας. το πώς είναι η ζωή στην περιφέρειά σας. Κοιτάμε σε περιφερειακό επίπεδο τι γίνεται. Σαρδινία. Βόρειος Ολλανδία. Νιουκάσιλ. Νότιος Δανία. Ρώμη. Στην Ιταλία. Μορέλος. Στο Μεξικό. Ή η εταιρική σχέση με την ΗΠΑ για τις ε, ε, βιώσιμες κοινότητες. Ορισμένα μόνο παραδείγματα κάποιων πολύ στοχευμένων περιφερειακών προσεγγίσεων σε ό,τι αφορά το πώς διαμορφώνεται η ζωή στην περιφέρεια του καθενός. Αντιλαμβανόμαστε ασφαλώς ότι αυτό που μετρά στις πιο πολλές ε, κοινωνίες ε, ξεπερνά το ΑΕΠ και το ΑΕΠ κατά κεφαλή. Προκειμένου να λάβουμε σωστές αποφάσεις για την πολιτική, δεν μπορούμε να κοιτάμε μόνο μόνο το οδόμετρο, θα πρέπει να κοιτάξουμε όλα τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Στον ΩΣΑ ε, δημιουργήσαμε λοιπόν ένα, μια ομάδα δικτών για να μας δείξει καλύτερα τι γίνεται. Και τώρα λοιπόν εστιαζόμαστε στις περιφέρειες, γιατί πιο πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν τη ζωή του κόσμου καθημερινά καθορίζονται σε τοπικό επίπεδο ουσιαστικά. Σας καλώ λοιπόν να, να ανακαλύψετε το website μας, το οποίο είναι διαδραστικό και επιτρέπει τη σύγκριση 362 περιφερειών σε 32 χώρες σε ό,τι αφορά 9 διαφορετικές διαστάσεις, σε ό,τι αφορά την ποιότητα ζωής. Για παράδειγμα, μπορείτε να δείτε τη σύγκριση Τοσκάνης και Τέξας στα θέματα υγείας. Σαξονία σε σχέση με το Κανθάι, όταν πρόκειται για θέματα ανεργίας υλικές ε, συνθήκες όπως πρόσβαση σε θέσεις εργασίας, ε, ε, μη υλικέ διαστάσεις, το περιβάλλον και το καθεξής. Όλα αυτά λαμβάνονται εξίσου υπόψη και πολλοί παράγοντες εξαρτώνται ουσιαστικά από το που ζει κανένας. Η εθνική μέση όρη ουσιαστικά δεν είναι καθοριστική, δεν μας λένε πολλά. Και τονίζουμε λοιπόν ότι θα πρέπει να δούμε πώς μεταφράζονται οι δημόσιες επενδύσεις σε ό,τι αφορά τι θέσει απασχόληση, τι ευκαιρίε, αυξάνοντα την ευημερία όλου του κόσμου. Και συχνά προσμετρούμε αυτό που μπορούμε εύκολα να καταμετρήσουμε. Για παράδειγμα, αριθμό κλινών στα νοσοκομεία. Αυτό είναι πολύ αντικειμενικό κριτήριο. Και πολύ αξιόπιστος δείκτης, αλλά αυτό δεν μας λέει φυσικά αν ο κόσμος είναι υγιής. Θα πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε διάφορους, ε, διάφορες διαστάσεις της ευημερίας για να επηρεαστεί ανάλογα και η σχετική πολιτική. Ε, η πιο καλή στόχευση λοιπόν των επενδύσεων για καλύτερα αποτελέσματα και πιο σωστή, σωστή επίδραση. Για παράδειγμα, το πρασίνισμα των υποδομών δεν έχει μόνο αποτελέσματα για το περιβάλλον, αλλά δημιουργεί και θέσεις ε, εργασίας, προωθεί κάποια είδη τεχνολογίας εκ παραλληλού. Όσο αυξάνονται λοιπόν σε έκταση τα αστικά κέντρα, η στοχευμένη επένδυση αποτελεί κάτι κρίσιμη σημασία, γιατί δύο από στους τρεις στις χώρες όσα μένουν σε πόλεις. Δεν χρειαζόμαστε λοιπόν διοικητικά εμπόδια. Αν καταφέρουμε να το πετύχουμε αυτό, ο κόσμος θα διαμορφωθεί διαφορετικός και γι' αυτό λοιπόν αναπτύξαμε μια μετροπολιτική, μετροπολιτική βάση δεδομένων 1.200 αστικές περιοχές βάσει κοινών ορισμών και κοινών μεθόδων. Και έτσι συμπεριλαμβάνεται μια μεγάλη ομάδα δεδομένων για τις 275 μεγαλύτερες πόλεις, οι οποίες φιλοξενούν παρεπιπτόντος το ίμιση του πληθυσμού του ΩΣΑ. Άρα έχει γίνει καλή καρτογράφηση. Και γι' αυτό οι συστάσεις που προέκυψαν από αυτές τις παρατηρήσεις και από τα γεγονότα αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Αυτή λοιπόν η δυτή προσέγγιση μας επιτρέπει να εξετάσουμε τι γίνεται μεταξύ αστικού χώρου και υπαίθρου. Οι μικρές κομμόπολεις και πόλεις όπως και οι μεγάλες πόλεις μπορούν να έχουν θετικό αντικτύπο σε όλη την περιφέρεια, μέχρι και 200 χιλιόμετρα πέρα από τα ωριά τους. Άρα δεν κοιτάμε μόνο τις πόλεις, αλλά και την οικονομική λεκάνη, την οικονομική περιφέρεια επιρροής των πόλεων αυτών. Και έτσι βλέπουμε ποιο είναι το χάσμα μεταξύ αστικού και χώρου και υπαίθρου, προκειμένου να μπορέσουμε να καλύψουμε το χάσμα αυτό μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε κάνει αναλύσεις και συστάσεις σε ό,τι αφορά τις ε, εταιρικές σχέσεις για την περιφερειακή ανάπτυξη μεταξύ πόλεων και υπαίθρου. Ένα βασικό θέμα είναι η γενική παραγωγικότητα στις πόλεις, αλλά υπάρχει και κόστος. Οι ε, μισθοί, για παράδειγμα, είναι πιο υψηλή, οι τιμές τείνουν να είναι πιο υψηλές στις πόλεις. Υπάρχει και μη νομισματικό κόστος, όπως για παράδειγμα η ρήπανση, ο χρόνος μεταφοράς προς την ε, εργασία. Όλα αυτά λοιπόν επηρεάζουν την ευημερία γενικά οι καλά οργανωμένες πόλεις μπορούν να μειώσουν σε κάποιο βαθμό αυτά τα αστικά μειονεκτήματα. Για παράδειγμα, οι πιο καλές δημόσιες συγκοινωνίες περιορίζουν τον χρόνο μεταφοράς και ε, περιορίζουν και την εκπομπή διοξυντή του άνθρακα. Και δίνουν και μεγαλύτερη πρόσβαση σε πιο πολλές θέσεις εργασίας στους πολιτές. Δυστυχώς, πολλές από τις πόλεις μας δεν μπορούν να πετύχουν αυτά τα πλέον εκτήματα. Και σε πολλές περιπτώσεις τα αστικά κέντρα ανταγωνίζονται τα μεν τα δεν και όχι δεν συνεργάζονται μεταξύ τους προκειμένου και έτσι τελικά τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι για να ξεπεράσουμε το μετροπολιτικό κατακριματισμό θα καταφέρουμε να πετύχουμε και καλύτερη περιβαλλοντική περιβαλλοντικές συνέπειες και μεγαλύτερη ικανοποίηση και των πολιτών. Πώς λοιπόν πρέπει να επενδύσουμε. σε ευρωπαϊκό τοπικό επίπεδο οι μεγάλες προκλήσεις είναι οι προεθνικές κυβερνήσεις που είναι πάνω από 90.000. Πολλές λοιπόν εξ αυτών ιδρύθηκαν σε διαφορετικές ε, εποχές, με πολύ διαφορετικές συνθήκες σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τη Γαλλία και τα σχετικά διαμερίσματα Ο κόσμος έχει αλλάξει έκτοτε. Ο πολιτικός ορισμός όμως εξακολουθεί να υφίσταται. Η οντότητα εξακολουθεί να υφίσταται. Πέρα από διάφορες συγχωνεύσεις, για παράδειγμα οι κομιτείες στη Σουηδία έχουν τα ίδια σύνορα που έχουν το 1634. Φυσικά δεν χρειάζεται να χαράξουμε εκ νέου του χάρτες μας, αλλά να σκεφτούμε κατά πόσο οι δομέ αυτές εξακολουθούν να είναι αποτελεσματικές και κατά πόσο ε, ταιριάζουν στη σημερινή πραγματικότητα σε ό,τι αφορά το 2014 περίπου το ίμιση των χωρών του ΩΣΑ εφαρμόσαν ή εφαρμόζουν κοινοτικές ε, νομαρχιακές ε, αλλαγές, μητροπολιτικές αλλαγές, προκειμένου να αναθεωρηθούν οι πολιτικές οντότητες μέσα στο ιστορικό της χώρας και αυτό αυτές οι μεταρρυθμίσεις σημαίνουν και μείωση των δαπανών. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτεί κάθε χώρα γιατί κάνει αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Θα πρέπει επίσης να σκεφτούμε πως οι κυβερνήσεις στα διάφορα επίπεδα και αυτό το διοικητικό συνοθήλευμα μπορούν να, μπορούν να αποφύγουν τις αλληλεπικαλύψεις και τα προσκόμματα και σε αυτό το, στις για το 2014 περιλαμβάνονται και συστάσεις για αποτελεσματικές δημόσιες επενδύσεις σε όλα τα επίπεδα των κυβερνήσεων. Αυτό είναι το βασικό εργαλείο του ΩΣΑ για να αντιμετωπιστεί το θέμα των ε, υποεθνικών κυβερνήσεων τάσει για αποτελεσματικές δημόσιες επενδύσεις σε όλα τα επίπεδα τοπικής και περιφερειακής κυβέρνησης. Τώρα, σε ό,τι αφορά συγκεκριμένε συγκεκριμένες ε, προκλήσεις, αναφέρουμε τρεις σε ό,τι αφορά το συντονισμό των κυβερνήσεων σε όλα τα διαφορετικά επίπεδα κυβερνήσεων και πολιτικών. Πώς μπορούν να ενισχύσουν τη δυνατότητα επενδύσεων και πώς μπορούν να πετύχουν το σωστό πλαίσιο για τις επενδύσεις. Χαιρόμαστε που η Επιτροπή των Περιφερειών επικύρωσε αυτές τις αρχές και ότι η τελευταία πολιτική συνοχή και οι σχετικέ ε, συμφωνίε εταιρική σχέση ε, επίση ε, συμπεριλαμβάνουν πολλέ από τι καλέ αυτέ πρακτικέ. Ελπίζω λοιπόν αυτέ οι δύο εκθέσει του ΩΣΑ να αποτελέσουν ωφέλιμα και χρήσιμα εργαλεία για τη δουλειά σα και να προωθήσουν την πιο δίκαιη και πιο πράσινη ανάπτυξη για να βελτιώσουν τη ζωή του κόσμου και την ευημερία των μελλοντικών γενναιών. Και σε αυτόν τον παγκοσμιοποιημένο κόσμο που ζούμε, οι πολίτες ε, απογοητεύονται όλο και πιο πολύ. Έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους και αισθάνονται χαμένοι όλο και πιο πολύ. Χάνουν την εμπιστοσύνη τους στους θεσμούς, σε όλα όσα έχουμε δημιουργήσει τα τελευταία 100 χρόνια. Υπουργοί, κοινοβούλια, πολιτικά κόμματα, πρωθυπουργοί, τραπεζικά συστήματα, πολυεθνικές. Άρα η συνεργασία μας καθίσταται όλο και πιο σημαντική προκειμένου να βοηθήσουμε τις κυβερνήσεις αλλά και τον κόσμο, τις κοινωνίες μας να αναπτύξουν καλύτερες πολιτικές για καλύτερη ζωή. Και θα ήθελα να τράξω την σημερινή ευκαιρία και να ευχαριστήσω τον Ιωάννης Χάν, να τον αποχαιρετήσω και να τον καλωσορίσω. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you. Thank you. Σας ευχαριστώ, Ευχαριστώ, κύριε Κουρία. Η επόμενη ομιλία μας είναι ένα μήνυμα το οποίο θα δοθεί μέσω ε, βίντεο από τον πρόεδρο κύριο Μπαρός. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, χαίρομαι που μπορώ να παίρνω το λόγο σε μια τόσο σημαντική ευκαιρία. Οι ημερίδες αυτές είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Κάποια από τα δίκτυα συνεργασίας που λειτουργήσαν επιτυχώς στην Ευρώπη προέρχονται από αυτές τις ανοιχτές μέρες, τις ημερίδες. Πολλά από τα προγράμματα έχουν επίσης ε, τις ρίζες τους στις ημερίδες αυτές και κάποιες από τις ιδέες οι οποίες περιλαμβάνονται στη νέα πολιτική μας προέρχονται από αυτήν την ετήσια συνάντηση. Την τελευταία δεκαετία συναντηθήκαμε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Οι χειρότερες οικονομικές, χρηματοπιστωτικές και κοινωνικές κρίσεις από την εκκίνηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης μας δοκίμασαν, αλλά παρά τις προβλέψεις πολλών επιβεβαιώσαμε ότι οι δυνάμεις της ολοκλήρωσης κυριάρχησαν μείναμε μαζί, μείναμε κοντά και στηρίξαμε ο ένας τον άλλον. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές διασώσαμε την ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Αυτό ήταν το σύνθημά μου. Και ε, οι, οι ηγέτες σε περιφερειακό επίπεδο ήταν οι καλύτεροι σύμμαχοί μας, έτσι ώστε να καλύψουμε τις απαιτήσεις ενός κόσμου που αλλάζει με πολύ μεγάλη ταχύτητα, πολύ ψηλή ταχύτητα αλληλεγγύη, υπευθυνότητα έχουν αρχίσει να δίνουν καρπούς. Έχουμε βάλει τα θεμέλια για μια σωστή και αηφόρο οικονομική ανάπτυξη. Είμαστε στο σωστό δρόμο, αλλά πρέπει να είμαστε ειλικρινεί. Ο δρόμος αυτός είναι μακρύς. Η πραγματικότητα είναι ότι η ανάκαμψη είναι αργή, άνηση και εύθραυστη και απειλείται επίσης από ό,τι φαίνεται και από γεωπολιτικές διαταραχές. Είναι κρίσιμο λοιπόν να μην αποκλίνουμε από την πορεία μας, να στηρίξουμε τις διαφορετικές μεταρρυθμίσεις για την ανταγωνιστικότητά μας στο μέλλον και τις θέσεις απασχόλησης. Δεν πρέπει να καθησυχάσουμε, ιδιαίτερα όταν τόσοι πολλοί ε, πολίτες, ιδιαίτερα νέοι πολίτες, αναζητούν τόσο πολύ καιρό να βρουν μια θέση απασχόλησης και καλύτερες συνθήκες ζωής και δείχνουν ορισμένοι ότι η Ευρώπη έχει αιμονή με τη λιτότητα. Εμείς όμως πρέπει να πούμε ότι βασικός στόχος μας είναι οι θέσεις απασχόλησης, οι καλές θέσεις απασχόλησης και καλύτερη ποιότητα ζωής για σήμερα και για αύριο. Αυτή είναι η στρατηγική του 2020. Κίνητρα για την ανάπτυξη. Κίνητρα για μια ευφυή ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς που να εδράζεται στην γνώση και την καινοτομία. Έχουμε πάρει και οδυνηρά μαθήματα από την κρίση στο παρελθόν. Μάθαμε σαν παράδειγμα ότι η ανάπτυξη όταν τροφοδοτείται από το χρέος, είτε το δημόσιο είτε το ιδιατικό είναι κάτι το τεχνικό και μία υφόρο. Γι' αυτό λοιπόν και η δημοσιονομική εξυγίανση και η χρηματοπιστωτική σταθερότητα είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την υγιή ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα. Η ιδέα μας όμως είναι πάντα η ανάπτυξη και παραμένει. Η επένδυση στην ανάπτυξη και στις θέσεις απασχόλησης του μέλλοντος μέσω της έρευνας και της καινοτομίας είναι ζωτικές. Γι' αυτό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντα είπαμε ξεκάθαρο ότι απαιτείται διαρθρωτική αλλαγή, αλλά ταυτόχρονα πέρα από τις μεταρρυθμίσεις απαιτούνται και επενδύσεις για το μέλλον. Αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπερασπίστηκε σκληρά τον προϋπολογισμό για τα επόμενα 7 χρόνια. Είναι ένας επενδυτικός, σύγχρονος προϋπολογισμός. Στοχεύει στην ανάπτυξη, στην απασχόληση και συμπληρώνει με σωστό τρόπο τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Εδράζεται στην ευρωπαϊκή διάσταση και δεν είναι υποκατάστατο των εθνικών προϋπολογισμών. Και ακριβώς επειδή η πολιτική συνοχής είναι το βασικό χρηματο... χρηματικό μέσο αυτής της δημοσιονομικής πολιτικής, θεωρούμε ότι πρέπει να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο την πολιτική συνοχής. Αλλάξαμε αυτήν την, αυτό το, το έθιμο αν θέλετε ή το συνήθιο των επιδοτήσεων που είχαμε και δώσαμε προτεραιότητα σε προγράμματα καινοτόμα, σε προγράμματα πράσινης οικονομίας και στην επίτευξη των στόχων της Ευρώπης του 2020. Δώσαμε δηλαδή μια λογική στις επενδύσεις μας και αυτή η νέα αντιμετώπιση οδήγησε στις εταιρικέ συμφωνίες με κάθε κράτος μέλος που ορίζουν μια στρατηγική η οποία θα, της οποίας θα επιδιωχθεί η εφαρμογή και ο καλύτερος τρόπος για την βελτίωση της χρηματοδότησης, γιατί το θέμα δεν είναι μόνο οι δαπάνες, είναι η ποιότητα των δαπανών, η ποιότητα της χρηματοδότησης. Όλα αυτά φυσικά δεν θα μπορούσαμε να τα πετύχουμε χωρίς την δική σας δραστήρια συμμετοχή. Είναι μια εξαιρετική ευθύνη αυτή βέβαια γιατί η πολιτική της συνοχής μπορεί πράγματι να κάνει πολλά για να βελτιώσει την καθημερινότητα των Ευρωπαίων, να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής και να δώσει ευκαιρίες απασχόλησης. Αυτό ακριβώς έχει σημασία για τους πολίτες μας. Αυτό ακριβώς έχει ε, σημασία γιατί δείχνει την προστιθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλληλεγγύη λοιπόν και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δώσαμε μάχη για τον προϋπολογισμό επενδυτικής φύσης. Αυτό δεν έχει στόχο τις Βρυξέλλες, έχει στόχο τις περιφέρειες, τα πανεπιστήμια, τους φοιτητές, τους ερευνητές, τους γεωργούς. Η πολιτική συνοχής λοιπόν δεν είναι μια παλιά πολιτική, είναι μια επενδυτική πολιτική και γνωρίζουμε ότι στην Ευρώπη αυτό που χρειαζόμαστε είναι οι επενδύσεις. Συνεπώς αγαπητοί φίλοι κατά τα τελευταία δέκα χρόνια Πράγματι βιώσαμε δραματικές στιγμές, εντατική πίεση. Αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι μπορούμε ξεκάθαρα να πούμε ότι αποδείξαμε την τεράστια ανθεκτικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντισταθήκαμε σε ισχυρότατες πιέσεις και όταν πολλοί προέβλεπαν το χειρότερο, δηλαδή την διάλυση της Ευρωζώνης ή ε, και τη διάλυση της Ένωσης μερικές φορές κάποιοι, εμείς δείξαμε ότι οι δυνάμεις της ολοκλήρωσης υπερίσχυσαν των δυνάμεων της πολυδιάσπασης. Και ακριβώς είναι συλλογική μας ευθύνη τα επόμενα δέκα χρόνια να είναι πιο λαμπρά. Και προσαρμοστήκαμε για να δείξουμε ότι είμαστε ισχυρότεροι και καλύτερα προπαρασκευασμένοι για τα προβλήματα και τις ευκαιρίες ενός κόσμου ε, που τρέχει με 100. Θέλω να σας ευχαριστήσω λοιπόν για τη στήριξή σας και για την επικοδομητική σας συνεργασία όλα αυτά τα πολύ δύσκολα και απαιτητικά χρόνια. Στις πιο δύσκολες στιγμές πάντα ήξερα ότι οι πολιτικοί ηγέτες σε όλα τα επίπεδα των περιφερειών, των πόλεων, ακριβώς επειδή έχουν την ευθύνη, κατανοούσαν και τις δύσκολες αποφάσεις τις οποίες χρειάστηκε να πάρουμε. Σας εύχομαι λοιπόν ό,τι καλύτερο, καρποφόρες συνεδριάσεις και ε, κυρίως εύχομαι κάθε επιτυχία για την περιφέρειά σας, της πόλης σας και το μέλλον της κοινή μας Ευρώπης. Ευχαριστώ. with Να συνεχίσουμε τώρα με τις δηλώσεις των Ευρωβουλευτών μελών της Επιτροπής ΕΡΕΤΖΙ και μελών της Επιτροπής των Περιφερειών. Να ξεκινήσουμε από την Επιτροπή των Περιφερειών, που είσαστε προσκεκλημένοι μας σήμερα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι το πρόγραμμα που έχουμε μπροστά μας μας αναγκάζει να ακούσουμε έναν από κάθε πολιτική ομάδα. Θα ξεκινήσουμε από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Schneider. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε. Μπορώ παρακαλώ να σας ζητήσω να μην μιλήσετε πάνω από δύο λεπτά ο καθένας από εσάς θα πάρει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Μου δώσατε 100% παραπάνω από όσο περίμενα. Το διπλάσιο μου δώσατε. Ήθελα να πω ότι ο χρόνος μας επιτρέπει μόνο μία μικρή πινελιά στον ε, σημερινό καμβά. Γι' αυτό θα ήθελα να κάνω μία γενική παρατήρηση. Ο τίτλος σήμερα είναι Growing Together, η αποκοινού ανάπτυξη. Αυτό είναι και λίγο αμφίσιμο όμως. Αφενός σημαίνει να να αναπτυχθούμε, να μεγαλώσουμε μαζί ή και να έχουμε κοινή ανάπτυξη, να γίνουμε ένα μετά. Και θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι είναι απαραίτητο για κάτι τέτοιο. με τη θέση του Επιτρόπου Χάν ότι για τα επόμενα χρόνια έχουμε θέσει πολύ καλές βάσεις στον τομέα της πολιτικής συνοχής επενδύσεις, ανάπτυξη, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, ε, δημιουργία ε, θέσεων απασχόλησης. Και έτσι θα μπορέσουμε ε, να συμβάλλουμε σε περισσότερη κοινή ανάπτυξη εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι πολύ σημαντική λειτουργία της κοινή πολιτικής συνοχής μας και θα ήθελα να επισημάνω ότι το πλαίσιο στο οποίο εργαζόμαστε σήμερα πολιτικά χρειαζόμαστε ακόμα περισσότερο αυτήν την αλληλεγγύη. Να αναφερθώ στην κρίση στην Ουκρανία που δεν είχαμε τις προηγούμενες δεκαετίες. Να αναφερθώ στην κατάσταση στην Μέση Ανατολή με το Ισλαμικό κράτος ε, να σας αναφέρω την κατάσταση στην ε, Βόρεια Αφρική, την ε, δραματική κατάσταση όσον αφορά την μετανάστευση, την, τους μετανάστες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό είναι σημαντικό να εργαστούμε μαζί και να αντιδράσουμε από κοινού σε αυτές τις προκλήσεις. Όλες αυτές οι γεωπολιτικές συγκρούσεις επηρεάζουν ε, και τις τοπικές ε, κοινότητες. Γι' αυτό μας συμφέρει να συμμετάσχουμε στην ε, διαδικασία λήψης αποφάσεων και γι' αυτό χαίρομαι που αποκοινούμε το Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βρισκόμαστε εδώ σήμερα στα Open Days που στο παρελθόν έχουν φανεί ιδιαίτερα χρήσιμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο σε μέλος της Επιτροπής Ρέτζη τον κύριο Τόμας Ντόιτς. Eh, Σας ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, αξιότιμοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Επιτρέψτε μου καταρχάς να εκφράσω την ευχαριστησή μου για το γεγονός ότι συνεχίζεται αυτή η καλή παράδοση σε ό,τι αφορά την διοργάνωση των ημερίδων αυτών σε συνεργασία με την Επιτροπή των Περιφερειών. Επιπλέον, το θέμα μας είναι να αναλύσουμε τις επιτυχίες και τα επιτεύγματα του τελευταίου καιρού και να επικεντρωθούμε σε αυτά και να αποφασίσουμε βάσει αυτών είναι, ποια θα είναι τα καθήκοντά μας ε, τα επόμενα χρόνια. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε τις ακροάσεις των υποψηφίων επιτρόπων. Οι ακροάσεις λοιπόν αυτές έλαβαν χώρα Και στο πλαίσιο αυτό η Επιτροπή Ρέτζι του Κοινοβουλίου έκανε ακρόαση στην υποψήφια Επίτροπο κυρία Κρέτου που θα είναι η υπεύθυνη και αρμόδια για θέματα περιφερειακής, ε, μάλλον πολιτικής συνοχής. Στην ακρόαση λοιπόν αυτή τονίστηκε επανειλημμένα ότι αποτελεί πρόβλημα το οποίο θα πρέπει, ότι υπάρχει ένα πρόβλημα κατεπήγων το οποίο θα πρέπει τάχιστα να επιλύσουμε. Το 2013 τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα έργα τα οποία έγιναν σε περιφερειακό επίπεδο και τα οποία ξεκίνησαν σε περιφερειακό επίπεδο περιλαμβάνουν ένα ποσό 23,4 δισεκατομμύρια τα οποία δεν έχουν αποπληρωθεί. Σε ό,τι αφορά δηλαδή εξελίξεις που έχουν ξεκινήσει αλλά όπου υπάρχει καθυστέρηση πληρωμών. Η καθυστέρηση πληρωμών λοιπόν αυτή ανέρχεται σε 23,2 δισεκατομμύρια. Αυτό σε αντίφαση με τους ισχύοντες κανόνες που ορίζουν ότι οι λαβαριασμοί αυτοί θα πρέπει να ελέγχονται μέσα σε 60 ημέρες και μετά να πληρώνονται. Αυτός ο κανόνας λοιπόν παραμελήθηκε. Και έτσι λοιπόν η περιφερειακή πολιτική χάνει την αξιοπιστία της πλέον. Η κυρία Κεωρκίεβα άλλη μια υποψήφια επίτροπος η οποία θα είναι αρμόδια για θέματα δημοσιονομικών στην επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μας ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια της ακρόασης της ότι αν συνεχιστεί αυτή η διαδικασία η καθυστέρηση πληρωμών στα τέλη του τρέχοντος έτου θα φτάσει τα 30-35 δισεκατομμύρια. Ελπίζω σε αυτές οι ημερίδες και εκείνη η περισυλλογή να μας βοηθήσουν όλους προκειμένου τα επόμενα χρόνια να μπορέσουμε να δισταθμίσουμε αυτά τα χρέη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έτσι να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη στην περιφερειακή πολιτική σε ό,τι αφορά δηλαδή τα έργα αυτά τα οποία μπορούν πραγματικά να χρηματοδοτηθούν και να καλυφθούν. Η χρηματοδότηση αυτή λοιπόν θα πρέπει να παρέχεται εγκαίρως από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα πρέπει πάντα να πληρώνονται λογαριασμοί. Και συνεχόμενη χρονική περίοδο, τα λειτουργικά προγράμματα θα πρέπει εγκαίρως και νομίμως να χρηματοδοτούνται. Ελπίζω λοιπόν να μπορέσουμε να αναλύσουμε καλύτερα τα πράγματα. Ευχαριστώ για την ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών. Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, κύριε Επίτροπε, κύριε Γενική Γραμματέα. Το τελευταίο την τελευταία μια μισή ώρα δεν ακούσαμε καμία λέξη πιο συχνά από τον όρο επενδύσεις. Ε, και πράγματι, εάν θέλουμε να ξεφύγουμε από την κρίση, χρειαζόμαστε έξυπνες επενδύσεις. Οι τοπικές αρχές ε, στην Ευρώπη καλούνται εδώ να παίξουν ιδιαίτερο ρόλο και γι' αυτό αποτελούν και σημαντική προτεραιότητα της πολιτικής μου ομάδας. Να φροντίσουμε δηλαδή η δυνατότητα επενδύσεων των τοπικών αρχών στην Ευρώπη όχι μόνο να διατηρηθεί αλλά να προωθηθεί. Η πρώτη αντιπρόεδρος ε, Μαρίνη έχει υποβάλει πρόταση ψηφίσματος ε, πριν ε, λίγο καιρό και περιλαμβάνεται εδώ η σύσταση του ΟΣΑ για τις δημόσιες επενδύσεις και νομίζω ότι Προσφέρεται έτσι μια σημαντική δυνατότητα συνεργασίας με τον ΩΣΑ. Το θέμα των επενδύσεων συνδέεται στενά με το νομοθετικό πλαίσιο στην Ευρώπη καθώς και τους κανόνες τους δημοσιονομικούς και την εφαρμογή τους στα κράτη-μέλη, διότι πολλές τοπικές αρχές αντιμετωπίζουν σημαντικά προγράμματα όσον αφορά τους λογιστικούς κανόνες και γι' αυτό συχνά αντιμετωπίζουν εμπόδια ε, στην ε, εφαρμογή ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Ο κύριος ε, Χάν είπε ότι έχουμε συνεργαστεί πολύ καλά τα τελευταία χρόνια. Αποτελεί λοιπόν πρόκληση αυτήν την συνεργασία να την επεκτείνουμε και σε άλλους τομείς της αρμοδιότητάς του και γι' αυτό πιστεύω ότι στον τομέα της πολιτικής γειτονίας, για παράδειγμα, ε, μπορούμε να εφαρμόσουμε την ε, τεχνογνωσία ε, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, για παράδειγμα, στην Ουκρανία ή στην διασυνοριακή συνεργασία. Πιστεύω ότι υπάρχουν δυνατότητες. Διότι έτσι μπορούμε να στηρίξουμε τις κυβερνήσεις Ουκρανίας και Μολδαβίας να δημιουργήσουμε ε, δυνατότητες ε, για τις ε, κυβερνήσεις τους για επενδύσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Κραέλ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να αναφερθώ σε αυτά που είπε ο προλαλής σας, ο συνάδελφος κύριος Λάμπερτς. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Χάν για την εξωτερική συνεργασία τα τελευταία πέντε χρόνια, καθώς και με την Επιτροπή των Περιφερειών. Πιστεύω ότι πραγματικά έχουμε ε, δημιουργήσει μια πολύ καλή πολιτική συνοχή, τουλάχιστον στο χαρτί. Τώρα αυτή η πολιτική θα πρέπει να εφαρμοστεί στις περιφέρειες και ελπίζω μέσα στην προσεχή εβδομάδα να μπορέσουμε να συζητήσουμε τα θέματα που μας ενδιαφέρουν. Αυτό που έχω συγκρατήσει εγώ και αυτό που θα είναι σημαντικό στην εφαρμογή των ε, προγραμμάτων ε, είναι το πώς θα γίνουν όλα αυτά στην πράξη. Θα ήθελα να αναφερθώ στην πολιτική γειτονίας. Είναι θετικά είναι θετικό το μήνυμα ότι ο Επίτροπος που μέχρι τώρα ήταν ε, αρμόδιος ε, για τις ε, περιφέρειες θα ασχοληθεί με το θέμα αυτό στο μέλλον. Πιστεύω ότι η περιφερειακή συνεργασία θα πρέπει να θέσει ένα σημαντικό παράδειγμα στον τομέα αυτόν. Σας εύχομαι καλή επιτυχία και ελπίζω στο μέλλον να μπορέσουμε να συνεργαστούμε και σε αυτόν τον τομέα πολιτικής. Έχω όμως ε, ένα επίγον ερώτημα. Θα ήθελα να δράξω την ευκαιρία να ρωτήσω πώς ρυθμίζονται οι πληρωμές. Πώς ως Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε στις ε, υποχρεώσεις ε, που έχουμε αναλάβει. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 23 δισεκατομμύρια ευρώ δεσμεύσεων ε, στα οποία δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε. Έχουμε μελλοντικά προγράμματα, αλλά δεν μπορούμε να πληρώσουμε αυτά για τα οποία ήδη έχουμε δεσμευτεί πολιτικά. Τι θα πούμε λοιπόν στις περιφέρειες τη στιγμή που δεν έχουμε χρήματα για αυτά που έχουμε υποσχεθεί Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό το μήνυμα που έχουμε να στείλουμε εδώ και θα χαιρόμουν εάν στις Open Days μπορέσουμε να στείλουμε ένα μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πληρώσει τα χρέη της στις περιφέρειες. Ευχαριστώ πολύ. Βερκέρκ. κύριος Βερκέρκ. Εξ ονόματος της, ομάδας των φιλελευθέρων, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω κυρία Μιχάλεμα που διοργανώνετε αυτή την ε, ημερίδα και τον Επιτροπό Χάν που ξαναθέτει το θέμα της αστικής ατζέντα. Να συγχαρώ επίσης τον κύριο Βαλκαρσέλ για την ε, εκλογή του ως Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είμαι βέβαιος ότι η φωνή των τοπικών και περιφερειακών αρχών θα ακουστεί στο Κοινοβουλίο. Θα ήθελα να πω ότι μου άρεσε η παρουσίαση του κυρίου Γενικού Γραμματέα, κυρίου Γκουρία, και στην ομιλία του ε, ήταν να επιβεβαιώνεται πολύ διάφορα θέματα τα οποία ανέφερα στην έκθεση μου για μια ενοποιημένη ευρωπαϊκή ατζέντα για τα αστικά κέντρα. Πρόκειται για ένα θέμα πάρα πολύ στις μόδας Πολλοί το συζητούν, οι πολιτικοί, οι επιστήμονες, οι ευθύνοντες. Ένα θέμα το οποίο όμως χρειάζεται πάρα πολύ να εφαρμοστεί στη σημερινή εποχή. Και μου άρεσε αυτό που είπε ο κύριος Γκουρία ό,τι αφορά το υποπεριφερειακό επίπεδο και το τι αποτελεί ε, περιφέρεια και πόλη. Είπατε ότι είναι η απόσταση που μπορεί να κάνει κανείς σε ένα άλογο. Η απόσταση που σήμερα μπορεί να καλύψει κανείς με ένα ποδήλατο σε μία μέρα. Αυτό νομίζω δίνει μια καλή διάσταση στην αστική συζήτηση και φυσικά χρειάζονται και τα κατάλληλα εργαλεία. Όλοι οι ομιλητές είπαν ότι χρειαζόμαστε πιο στοχευμένους πόρους για να βοηθήσουμε την οικονομία σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Τα κράτη-έθνη είναι πολύ μακριά από τον τόπο για να γνωρίζουν τι χρειάζεται και τι αποδίδει. Και χρειάζεται λοιπόν τα εργαλεία του ΩΣΑ να μας βοηθήσουν για να κατανοήσουμε καλύτερα το τι συμβαίνει στην κάθε περιφέρεια και προκειμένου να είμαστε όσο πιο αποτελεσματικοί γίνεται με τις κατευθυντήριες γραμμές που έχουν και σε ό,τι αφορά την διοργάνωση των δημοσίων πόρων. Προσβλέπω στη συνεργασία με όλους σας, προκειμένου αυτό να καταστεί η αλήθεια για την καλύτερη μελλοντική Ευρώπη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει η Πρόεδρος, και τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Τόμασίτσου από το ECR, Συντηρητική και Μεταρρυθμιστές. Ευχαριστώ πολύ. Η πολιτική συνοχή αποτελεί το βασικό επενδυτικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελεί πάνω από το 1 τρίτο του προϋπολογισμού. 150 δισεκατομμύρια ευρώ είχαμε σε τέτοιες επενδύσεις σε τελευταίο καιρό. Είναι σημαντικό λοιπόν να προσαρμοστούν τα σχετικά προγράμματα προκειμένου να εφαρμοστούν και οι στόχοι για την Ευρώπη του 2014 Κάθε περιφέρεια λοιπόν πρέπει να αναπτύξει τα πλανεκτήματά της προκειμένου να έχουμε και σωστή επένδυση στους τομείς οι οποίοι είναι πολλά υποσχόμενοι σήμερα. Αυτό τι σημαίνει ότι θα πρέπει να ορίσουμε και στόχους προσμετρήσιμους, καταμετρήσιμους και θα πρέπει λοιπόν να θέσουμε στόχους ποσοτικοποιημένους προκειμένου στη συνέχεια να μπορέσουμε να κρίνουμε κατά πόσον οι επενδύσεις ε, ε, προώθησαν την απασχόληση και την ανάπτυξη στην Ευρώπη κάθε ευρώ που δαπανάτε θα πρέπει να έχει το μέγιστο δυνατό αντίκτυπο σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα. Από τις περιφέρειες λοιπόν περιμένουμε να δραστηριοποιηθούν ενεργά στη διαμόρφωση των προγραμμάτων αυτών προκειμένου η πολιτική συνοχή να στεφτεί με επιτυχία πραγματικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Σίλμπερκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριοι και κυρίες Ευρωβουλευτές, κύριε Επίτροπε, καταρχάς θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Χάν και τον Γενικό Γραμματέα του ΟΣΑ, τον κύριο Γκαρία, στην ενακτήρια αυτή σύνοδο των Open Days. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα επίσης να σας συγχαρώ για το νέο διορισμό σας ως Επιτρόπου και θα ήθελα να πω ότι πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να σημειώσει τις συστάσεις του ΟΣΑ για την μεγαλύτερη ολοκλήρωση μεταξύ των διαφόρων πολιτικών τομέων, όπως είναι η γεωργία, η περιφερική πολιτική και άλλες. Έχω Επίσης, μια ερώτηση προς τον Όσα Ο ΩΣΑ έχει κάνει έρευνες ε, σχετικά με τις ε, σχέσεις μεταξύ των ε, διαφόρων υπαίθριων περιοχών. Έχουν κάνει πολιτική ανάλυση σχετικά με τις επενδύσεις στις υπαίθριες περιοχές. και για τις αστικές περιοχές. Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις επενδύσεων στην απασχόληση και την ανάπτυξη σε αγροτικές περιοχές ε, σύμφωνα με τις αναλύσεις του ΩΣΑ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τον λόγο στον κύριο Γιάκοφτσης ε, της ομάδας ALDE της ε, Επιτροπής ΡΕΤΖΙ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι εκ μέρους των μελών ε, της ΑΛΔΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ήθελα να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλους τους συναδέρφους μας στην ε, Επιτροπή των Περιφερειών. Ήμουν ε, συνειδητής κατά κάποιο τρόπο των Open Days πριν από 10-12 χρόνια και ως ε, Ρία, είχα τη δυνατότητα να συμμετάσχω τότε στις Open Days. Γνωρίζω πόσο σημαντική είναι η εκδήλωση αυτή για την πολιτική συνοχή και για τη δημοκρατία. Θα ήθελα να συμφωνήσω με τις ανησυχίες των συναδέλφων μας ε, από το ΕΛΚ και τους σοσιαλιστές και δημοκράτες που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση ή μάλλον την ελληπή χρηματοδότηση των προγραμμάτων που έχουν εγκριθεί και εφαρμοστεί. Είναι πολύ σημαντική αυτή η ανησυχία. Εκ μέρους της ΑΛΤΕ θα ήθελα να καλέσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλους όσους πρέπει να λύσουν το πρόβλημα αυτό να το κάνουν όσο γίνεται πιο σύντομα. Διότι υπάρχουν σημαντικές ανησυχίες μεταξύ των εταίρων μας σε όλη την Ευρώπη. Σήμερα θα ήθελα να τονίσω ένα θέμα τελείως διαφορετικό. Εδώ και αρκετό καιρό σκέφτομαι ποια είναι τα προβλήματα απορρόφησης ε, κατά την εφαρμογή των διαφόρων προγραμμάτων και γιατί τόσες χώρες στην Ευρώπη δεν καταφέρνουν να διοχετεύσουν ε, τα χρήματα αυτά στις περιφέρειες και στις πόλεις. Θα ήταν πολύ χρήσιμο κάτι τέτοιο να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στις περιφέρειες όπου εφαρμόζονται τα προγράμματα θα ήταν χρήσιμο να υπάρχει μια task force, μια ειδική ομάδα για την ενίσχυση της δυνατότητας απορρόφησης σε διαφόρων κρατών και περιφερειών. Στο πλαίσιο αυτό πιστεύω ότι όλοι θα πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες, διότι είμαι πεπισμένος ότι οι πολίτες που Ε, μαθαίνουν ότι ε, δεν ε, χρησιμοποιούνται οι πόροι αυτοί, δεν θα θεωρήσουν χρήσιμη την πολιτική αυτή, διότι δεν διοχετεύονται τα χρήματα εκεί που υπάρχουν οι μεγαλύτερες ανάγκες. Θα ήθελα επίσης να προτείνω στον νέο Επίτροπο να έχει ένα σύστημα να δημιουργήσει ένα σύστημα διαχείρισης των κρίσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σκιμόρ. Um, e- Σας ευχαριστώ. Από πλευράς της, Επιτροπής ομάδας ECR θα ήθελα να καλωσορίσω τη συζήτηση αυτή. Ο κύριος Γκουρία μίλησε για σημαντικούς τομείς όπως η πιο στενή συνεργασία. Θα ήθελα να αναφέρω τρεις τομείς όπου η ομάδα του ECR πιστεύει ότι πρέπει να επικεντρωθούμε πιο πολύ. Καταρχάς, να εξετάσουμε πιο πολύ τα θέματα προσβασιμότητας σε, θέματα, σε, σε ό,τι αφορά τις ε, περιοχές που έχουν ε, μια ενεκτική πρόσβαση σε ό,τι αφορά τις ορεινές περιοχές για παράδειγμα ή τις εξοχος απόκεντρες περιοχές. Θα πρέπει να κοιτάξουμε το σύνολο των περιφερειών σε ό,τι αφορά τον σχεδιασμό και οι περιφέρειες αυτές ε, δεν θεωρούνται ακόμα ως κοινή ευρωπαϊκή πρόκληση. Καλούμε λοιπόν την νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δημοσιεύσει μία πράσινη βίβλο για το θέμα αυτό, προκειμένου το θέμα αυτό να συζητηθεί από τους εμπλεκόμενους φορείς και από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να υπάρξει και η σωστή ανταπόκριση. Κατά δεύτερον, να υπάρξει ανθεκτικότητα σε κρίσεις και καταστροφές θα πρέπει να βρούμε μια προσέγγιση για την ανάκαμψη προκειμένου να αναπτύξουμε περαιτέρω την ετοιμότητά μας και την ανθεκτικότητά μας. Και τέλος θα πρέπει να επικεντρωθούμε στη μείωση της γραφειοκρατίας και τη μείωση των γραφειοκρατικών εμποδίων. Αυτό όχι μόνο θα αυξήσει την διεθνή μας ανταγωνιστικότητα και αποτελεσματικότητα, αλλά και τις δυνατότητες απορρόφησης των ταμείων, των πόρων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Μπράνις Ρόπε. Σας ευχαριστώ. Εγώ είμαι καινούργια μέλος εδώ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πριν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήμουν δήμαρχος επί 22 έτη και ξέρω πραγματικά λοιπόν τι σημαίνει και τι μπορούν να κάνουν οι τοπικές και περιφερειακές αρχές για τους πολίτες μας. Γι' αυτό λοιπόν ιδιαίτερος ε, χάρηκα σήμερα για το γεγονός ότι μπορώ να σας το λόγο εξ ονόματος της ομάδας της ΓΚΟΕ. Η Ευρώπη ξεκινάει από τους πολίτες της. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι ο τίτλος της ημερίδας «Η έξυπνη ευφυή επένδυση για τον κόσμο» είναι πάρα πολύ επίκαιρη γιατί θα πρέπει να ξεπεράσουμε την κρίση, να δώσουμε όθηση στην αγωνιστικότητά μας. Πιστεύω ότι όλες οι αρχές τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης στην Ευρώπη κατανοούν ότι η ανταγωνιστικότητα και η ποιότητα ζωής σε όλη την Ευρώπη δεν θα επιτευχθούν ποτέ χωρίς να υπάρχει πολιτική συνοχή σωστά εφαρμοσμένη. Οι αρχές περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης αποτελούν πολύ σημαντικό παράγοντα γιατί είναι ο πιο κοντινός παράγοντας στους πολίτες. Και γι' αυτό λοιπόν η Επιτροπή των Περιφερειών εξακολουθεί να συμβάλλει στην βελτίωση της πολιτικής συνοχής. Εμείς στην ομάδα μας δε θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να διασφαλίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει αποτελέσματα σε ό,τι αφορά την πολιτική συνοχή για το όφελο όλων των πολιτών. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Ντεμάτο. E για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η ανάπτυξή τους συνδέεται άμεσα και πάντα με την εξέλιξη μιας περιοχής, μιας συγκεκριμένης περιφέρειας. Για να είναι πραγματικά βιώσιμες και οικονομικά και ε, περιβαλλοντικά, είναι απαραίτητο να τις φροντίσουμε. Έχουμε κάποιες πόλεις μπροστά μας και κάποιες περιφέρειες οι οποίες ήταν θα έλεγε κανείς μόνο βιομηχανικές σε τεράστιες διαστάσεις και που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα πλέον σε επίπεδο αηφορίας και ανάπτυξης. Απαιτείται λοιπόν συνεργασία ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και την Επιτροπή των Περιφερειών. Είμαστε διαθέσιμοι να συνεργαστούμε. Thank you. Thank you very Σας ευχαριστώ πολύ. φτάνουμε στα συμπεράσματα και θα δώσω το λόγο στον κύριο Βαλκάρ Σελσίσο από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Δεν νομίζω ότι έτσι και αλλιώς ε, χρειάζονται στην παρούσα φάση συμπεράσματα, έτσι κι αλλιώς έπεται η μεικτή συνεδρίαση των δύο επιτροπών, του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής των Περιφερειών. Να σας ευχαριστήσω όλους για την παρουσία σας εδώ, για την έναρξη το σημερίδας για το 2014. Ελπίζω να πάνε τα πράγματα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το τεχνικό περιεχόμενο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το θέμα είναι όμως ότι πρέπει να είναι σημαντική και η συνάντησή μας σε προσωπικό επίπεδο για να μπορέσουμε να ανταλλάξουμε πρακτικές και ιδέες έτσι ώστε τα επόμενα 7 έτη στην περιοχή της περιφερειακής πολιτικής και της συνοχής να στεφθούν από επιτυχία για την Ευρώπη, γιατί αυτό θα βοηθήσει τους πολίτες, τίποτα άλλο. Thank you. Thank you, Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε. Τώρα, για τα πραγματικά συμπεράσματα θα δώσω το λόγο στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής των Περιφερειών, τον πρώτο Αντιπρόεδρο της Επιτροπής των Περιφερειών, την κυρία Μαρίνη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ όλους για τη συνεισφορά σας στην συζήτηση. Να ευχαριστήσω τον Επίτροπο, τις Προέδρους, και τους Προέδρους των Επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής των Περιφορίων. Εδώ και 12 χρόνια οι ημερίδες αυτές είναι καθοριστική στιγμή για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές. Πρωταγωνιστούμε σε μια στιγμή διαλόγου και αντιπαράθεσης με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά όργανα. Προβαίνουμε σε ανταλλαγή χρηστών πρακτικών και ταυτόχρονα η φετινή συνάντηση θα πρέπει να αντιμετωπίσει σοβαρά το θέμα της αύξησης των δυνατοτήτων αύξησης των ευφυών μορφών επένδυσης που θα δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης, θα δημιουργήσουν ανάπτυξη. Αλλά όπως είπα θα πρέπει να βελτιώσουν και την ποιότητα της ζωής των πολιτών. Γι' αυτό είναι ευφυείς μορφές ε, ε, ε, επένδυσης απαιτούνται. Βρισκόμαστε στην αρχή, στη νέα περίοδο προγραμματισμού της πολιτικής συνοχής από το 2014 μέχρι το 2020 και γι' αυτό από την πλευρά των περιφερειακών και τοπικών αρχών να πούμε ότι η πολιτική συνοχή είναι ένα από τα βασικά μέσα. Σε μερικές περιοχές είναι το μοναδικό μέσο που έχουν στη διάθεσή τους οι τοπικές αρχές έτσι ώστε να μειώσουν τις διαφορές των περιφερειών μεταξύ τους, αλλά ταυτόχρονα να μειώσουν και τις διαφορές στην ανάπτυξη στο εσωτερικό των ιδίων αυτών των περιφερειών και έτσι να βελτιώσουν την ζωή των πολιτών. Νομίζω λοιπόν συμπερασματικά τρία πράγματα πρέπει να πούμε. Πρώτον να αναφερθώ στη συνεισφορά του Γενικού Γραμματέα του ΟΣΑ Αναφέρθηκε στην ανάγκη να χρησιμοποιήσουμε ένα επιπλέον μέσο του ΑΕΠ έτσι ώστε πέραν του ΑΕΠ για να προσμετρήσουμε όχι μόνο τους ρυθμούς ανάπτυξης αλλά και την αίσθηση ευημερία που έχουν οι πολίτες. Κάποια στιγμή πιστέψαμε ότι το ΑΕΠ μετράει τα πάντα και ξεχάσαμε τα υπόλοιπα τα οποία κάνουν τη ζωή άξια να τη ζει κανείς. Γι' αυτό λοιπόν προς την κατεύθυνση αυτή τώρα κάνουμε κάποια σωστά βήματα. Η Επιτροπή των Περιφερειών συνεισέφερε και αυτή από την πλευρά της τα τελευταία χρόνια για την προσμέτρηση της προόδου όχι μόνο με το ΑΕΠ αλλά και με άλλες πολιτικές. Υπάρχει και η έκθεση Βόσνιακ του Προέδρου της ΚΟΤΕΡ, της Επιτροπής ΚΟΤΕΡ για τα αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής μετά το 2013. Έχουμε λοιπόν ανάγκη και από δείκτες διευρυμένους, οι οποίοι να προσμετρούν την πρόοδο και μέσω άλλων χαρακτηριστικών. Έχουμε επίσης ανάγκη να σκεφτούμε προσεκτικά το τι συνέβη το 2008-2013. 20% λιγότερες πραγματικές σε πραγματικούς αριθμούς επενδύσεις δημόσιες. Η κρίση δηλαδή μείωσε συστηματικά τις δημόσιες επενδύσεις και όπως περιλαμβάνεται και στην έκτη έκθεση για την συνοχή, εάν εμείς δεν λάβουμε υπόψη την μείωση των διαφορετικών ποσών, τότε αυτή η μείωση ε, μπορεί να γίνει ακόμα περισσότερο δραματική. Η πολιτική λοιπόν, η ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής αυτά τα χρόνια της κρίσης, παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, ήταν ένας από τους πιο σημαντικούς τρόπους δημοσίων επενδύσεων στη διάθεση των τοπικών και περιφερειακών αρχών. Οι σημερινές εργασίες λοιπόν και οι παρεμβάσεις τις οποίες ακούσαμε κατά τη διάρκεια του πρώτου τμήματος αυτού των εργασιών και αυτά που θα ακούσουμε στη συνέχεια, από πλευρά τη Περιφερειακή Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη Επιτροπή Κοτέρ τη Επιτροπή των Περιφερειών θα δείξουν και το επίπεδο λειτουργικότητα τη επομένη ε, ε, προγραμματική περίοδου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει κάνει μια πρόταση την οποία συμμεριζόμεθα εμεί να ευνοήσουμε όσο περισσότερο γίνεται την σωστή δαπάνη ε, των διαφθορτικών ταμείων προς συγκεκριμένα προγράμματα κάνοντας ό,τι μπορούμε έτσι ώστε τα διαρθρωτικά αυτά μία να χρησιμοποιούνται με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα. Έτσι ώστε, σαν παράδειγμα, τα προβλήματα συγχρηματοδότησης των διαρθρωτικών ταμείων και σε περιφερειακό επίπεδο και σε κοινωνικό επίπεδο και σε επίπεδο τοπικών και περιφερειακών αρχών θα πρέπει να θεωρούνται εκτός ε, των κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας. Με τον τρόπο αυτό θα ξεμπλοκάρουμε τα μεγάλα έργα, τα απαραίτητα για την ανάπτυξη, τα οποία προς το παρόν προχωρούν με πολύ αργή ταχύτητα. Λοιπόν, δεν είναι συμπέρασμα ίσως, είναι ευχή, αλλά πρέπει η συνάντηση αυτή να βελτιώσει την ποιότητα απορρόφησης των διαρθρωτικών πιστώσεων και να δώσει κίνητρα στις τοπικές αρχές να ενισχύσουν ε, τις επενδύσεις αυτές που θα βελτιώσουν με τη σειρά τους την ποιότητα της ζωής των πολιτών. Thank you. Σας ευχαριστώ. Αυτή ήταν η καταληκτική ομιλία σε ό,τι αφορά την ενακτήρια αυτή συνεδρίαση των ημερίδων του 2014. Και τώρα θα συνεχίσουμε με την κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής Ρέτζι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής Κοτέρ, Επιτροπή Περιφερειακής ε, Πολιτικής Συνοχής της Επιτροπής των Περιφερειών. Θα παρακαλέσω τους ομιλητές να λάβουν θέσεις. Ladies and gentlemen, please. Κυρίες και κύριοι, σας παρακαλώ καθίστε. Θα συνεχίσουμε με την κοινή συνεδρίαση των επιτροπών μας. May we begin? Μπορούμε παρακαλώ να ξεκινήσουμε. I'll ask all the members of the committees to take their... Καλό τα μέλη των επιτροπών να καθίσουν. Meeting of the committees. Thank you. Κύριε Βόσνιακ, μέλη της Επιτροπής ε, ΚΟΤΕΡ, της Επιτροπής των Περιφερειών και αγαπητοί συνάδελφοι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι, χαίρομαι που μπορώ σήμερα να σας καλωσορίσω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι πρώτη φορά που η κοινή μας συνεδρίαση γίνεται ε, σε αυτήν την αίθουσα και ελπίζω η συνεδρίασή μας σήμερα να αποτελέσει ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις και να ξεκινήσουμε μια επικοδομητική συζήτηση πάνω σε κοινού τομεί δράση. Κατά τη διάρκεια της φάσης διαπραγματεύσεων ε, του νομοθετικού πακέτου για την πολιτική συνοχή 2014-2020, η Επιτροπή μας επωφελήθηκε πάρα πολύ από τις συμβουλές και τις εμπειρίες των συναδέρφων μας στην ΚΟΤΕΡ. Προσβλέπουμε στις ε, συνεισφορές σας κατά την φάση εφαρμογής. Ιδιαίτερα προσλέπουμε στην γνωμοδότησή σας πάνω στην έκτη έκθεση συνοχής. Γνωρίζω τις προσδοκίες που έχετε περιγράψει στο ψήφισμα της Επιτροπής των Περιφερειών του Ιουνίου του 2014 για την ε, νέα νομοθετική θητεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι επενδύσεις ε, στις στους Δήμους της Ευρώπης για περισσότερες ε, θέσεις απασχόλησης σε ανάπτυξη και βιωσιμότητα είναι απαραίτητες ε, για να διασφαλίσουν ε, την προετοιμασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις προκλήσεις του μέλλοντος. Την επόμενη χρονιά η Επιτροπή Ρέτζι θα επικεντρωθεί στην ε, έκτη έκθεση ε, οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής ε, συνοχής στην αστική διάσταση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ανάπτυξη κατευθυντηρίων γραμμών πάνω σε μέτρα που σχετίζουν που συσχετίζουν την αποτελεσματικότητα των επενδυτικών και διαρθρωτικών ταμείων με την καλή οικονομική διακυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την ε, Αδριατική και το Ιόνιο. Κυρίες και κύριοι, θέλουμε να δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τα εργαλεία της πολιτικής συνοχής. Αυτή η συζήτηση είναι ιδιαίτερα επίκαιρη. Η επόμενη προγραμματική περίοδος ε, περιμένουμε να είναι μια από τις πιο δύσκολες εδώ και πολλά χρόνια. Μια δεκαετία ε, οικονομικής κρίσης έχει πληγώσει πολλές από τις περιφέρειές μας ε, και είναι απαραίτητο τα Ευρωπαϊκά Ταμεία να παρουσιάσουν αποτελέσματα όσο γρήγορα και όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται. Γνωρίζουμε ότι ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, για την περιφερειακή πολιτική συχνά έχει υποστεί κριτική και περιμένουμε ε, αυξημένο δημόσιο έλεγχο σχετικά με το πώ χρησιμοποιούνται τα περιφερειακά ταμεία. Θα πρέπει να διατηρήσουμε τι δεσμεύσει μα στην ενδιάμεση αναθεώρηση του πολιτού ε, δημοσιονομικού πλαισίου και είναι καθήκον μας να παρουσιάσουμε τα μέγιστα αποτελέσματα για την ανάπτυξη και την δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην Ευρώπη. Οι περιφέρειες και οι πόλεις ε, είναι κεντρικοί παράγοντες ε, στην εφαρμογή πολιτικής. Ευτυχώ έχουμε νέα και αποτελεσματικά εργαλεία συμπεριλαμβανομένων των ολοκληρωμένων εδαφικών επενδύσεων ε, και ε, της ε, τοπικής ανάπτυξη, που λαμβάνει κατευθύνσει από τις ίδιε τι κοινότητε. Οι τοπικές κοινότητε θα παίξουν κεντρικό ρόλο στην παρουσίαση αποτελεσμάτων μέσω αυτών των εργαλείων και μια τοπική προσέγγιση είναι ένα χαρακτηριστικό κλειδί της νέας πολιτικής και θα πρέπει να εφαρμοστεί με την αυξημένη συνεργασία μας οι Επιτροπές Ρέτζι και Κοτέρ μπορούν να βοηθήσουν τις περιφέρειες και τις πόλεις ε, στη διαδικασία αυτή. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και ελπίζω να έχουμε επικοδομητική ανταλλαγή απόψεων στη σημερινή συνεδρία. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Αγαπητά μέλη τη Επιτροπή Ρέτζη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αγαπητοί συνάδελφοι τη Επιτροπή των Περιφερειών, κυρίε και κύριοι, είμαι πολύ χαρούμενο που βρισκόμαστε λοιπόν όλοι εδώ σήμερα για την κοινή αυτή συνεδρίαση τη Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ε, Περιφερειακή Ανάπτυξη και τη ε, Επιτροπή τη Επιτροπή των Περιφερειών για την ε, πολιτική περιφερειακή συνοχή. Είναι η πρώτη φορά που αυτή η εκδήλωση λαμβάνει η χώρα στο ημικύκλιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά μάλιστα κατευθείαν από την επίσημη, το επίσημη κίνηση των ημερίδων. Ευχαριστώ ιδιαίτερα στην κυρία Μιχαήλοβα και την ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχουν, μας έδωσαν αυτή την ευκαιρία. Θα ήθελα να μιλήσω τώρα πολωνικά κυρίες και κύριοι. Κυρίες και κύριοι, οι κοινέ συνεδριάσεις Επιτροπή Ρέτζη και Κοτέρ πάντα ήταν μια καλή ευκαιρία για σωστή ανταλλαγή απόψεων. Θα ήθελα να καλωσορίσω τα νέα μέλη της Επιτροπής Ρέτζη και να χαιρετήσω εκείνους τους οποίους γνωρίζουμε και με τους οποίους είχαμε πολλές ευκαιρίες να συνεργαστούμε κατά το παρελθόν για το πακέτο της συνοχής. Στην παρούσα φάση Βρισκόμαστε στην πιο κρίσιμη φάση των διαπραγματεύσεων για θέματα εταιρικής σχέσης με πολλές χώρες, καλό, καθώς και σε ό,τι αφορά πολλά λειτουργικά προγράμματα σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Έχουμε πολλές ε, προσδοκίες σε ό,τι αφορά τις χρηματοοικονομικές προοπτικές και οι προσδοκίες αυτές συνδέονται με την βέλτιστη αξιοποίηση των δημοσιονομικών πόρων που μας διατίθενται εκ παραλλήλου, αντιλαμβανόμαστε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δυστυχώς έχει εισαγάγει πολύ αυστηρούς κανόνες για την διαχείριση των κονδυλίων αυτών και θα πρέπει να τονίσουμε ότι ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα τα καινούργια εργαλεία και μέσα τα οποία εισήχθησαν και θα δώσουν την δυνατότητα να εφαρμοστεί καλύτερη αστική πολιτική. Θυμόμαστε την ε, έκθεση για τις πόλεις του μέλλοντος που περιγράφει με πολύ σωστό τρόπο τις προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζουν και πρόκειται να αντιμετωπίσουν στα επόμενα χρόνια οι πόλεις καθώς και τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να εισαχθούν προκειμένου να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις αυτές. Οι ενοποιημένες εδαφικές επενδύσεις αποτελούν το εργαλείο για να συνενωθούν οι διάφοροι εμπλεκόμενοι φορείς. Ένα εργαλείο το οποίο θα πρέπει να λειτουργήσει ως κίνητρο για την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Αλλά έτσι αναπτύσσεται και μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση των πόρων για την ε, εδαφική ανάπτυξη σε πολλά τοπικά προγράμματα χρησιμοποιούνται κάποια μέσα για την ενεργοποίηση των τοπικών επιχειρήσεων. Μια τοπική ανάπτυξη, πνοή ανάπτυξης, η οποία προέρχεται από τις τοπικές κοινότητες. Και αυτή η τοπική ανάπτυξη υπό την αιγίδα των τοπικών κοινωνιών είναι πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο, το CLLD. Στην Ευρωπαϊκή Έπειρο, λοιπόν, είναι πολύ διαφορετικές εντυπώσεις που επικρατούν για τις διαπραγματεύσεις αυτές. Σε ορισμένες περιπτώσεις φαίνεται ότι μας φαίνεται πάρα πολύ δύσκολη η διαπραγμάτευση γιατί τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιφερειάς μας θεωρούμε ότι δεν έχουν ληφθεί υπόψη. Από την άλλη, θεωρώ ότι έχουμε την, το δικαίωμα να αμφισβητούμε τα ζητήματα τα οποία άλλωστε τύχθησαν και εδώ σήμερα. Και θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να τα συζητήσουμε όλα αυτά, να υπάρχει δυνατότητα συζήτηση εκ παραλλήλου, να αντιλαμβανόμαστε ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να καταχραστούμε, να χρησιμοποιήσουμε με λάθος τρόπο τα κονδύλια αυτά. Αυτό είναι προφανές και εγώ προσωπικά θεωρώ ότι η μεταφορά της τεχνολογίας και η μεταφορά από την επιστήμη στην τεχνολογία στην, επιστήμη, στην ε, οικονομία αποτελεί ένα πάρα πολύ κέριο ζήτημα δεδομένων και των συνθήκων που επικρατούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναρωτιέμαι κατά πόσον μπορούμε με δέοντα τρόπο να διαχειριστούμε και τα κονδύλια αλλά και την ε, όλη διαδικασία. Ιδιαιτέρως ε, ανησυχώ και για τις αφόρμητες αντιδράσεις από πλευράς των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων. Πιστεύω ότι όταν έχουν εκχωρηθεί κάποια κονδύλια για την πολιτική συνοχής, δεν θα πρέπει να γίνεται αναδιανομή των πόρων αυτών. Θα πρέπει συγκεκριμένα να χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της πολιτικής συνοχής. Και ίσως ε, να πρέπει να γίνουν κάποιες διορθώσεις, κάποιες τροποποίησεις, αλλά από πλευράς ε, τοπικών και περιφερειακών αρχών θα πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες προκειμένου αυτές οι διορθώσεις να μην είναι απαραίτητες. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία κυρίες και κύριοι να ανταλλάξουμε απόψεις. Έως τώρα συζητήσαμε τη μορφή των πολιτικών μας και των στρατηγικών μας σε ό,τι αφορά τους συγκεκριμένους κανονισμούς. Οι συζητήσεις αυτές σε πολλές περιπτώσεις είναι δύσκολες και χρονοβόρες, αλλά σήμερα θα πρέπει να συζητήσουμε το πώς θα εφαρμοστούν πλέον αυτές οι πολιτικές και πιστεύω ότι θα πρέπει να αναρωτηθούμε πώς αυτά τα νέα εργαλεία, αυτά τα νέα μέσα θα λειτουργήσουν στα διάφορα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιοι είναι οι όροι και οι συνθήκες που προαπαιτούνται προκειμένου να σταθεί με επιτυχία αυτή η πολιτική συνοχή. Πώς οι αρχέ τοπική και περιφερειακής αυτοδιοίκησης μπορούν να ασκήσουν πολιτική και εξουσία για να είναι ομαλή αυτή η διαδικασία. Σε ποιο βαθμό έχει απλοποιηθεί ή έχει επιπλακεί αυτή η διαδικασία, αυτές οι προδιαγραφές εξάντες προφανώς θα επηρεάσουν και την αποτελεσματικότητα αλλά και την ταχύτητα των έργων. Και τέλος, θεωρώ ότι θα πρέπει να αναρωτηθούμε για θέματα εφαρμογής. Η εμπειρία μας ε, καταδεικνύει ότι είναι πολύ διαφορετική η ιστορία της κάθε χώρας. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να διευκολύνουμε τη διαδικασία αυτή και την... Ε, σε ό,τι αφορά τις αιτήσει. Έχουμε καθυστέρηση 45 λεπτών κυρίε και κύριοι, αλλά θεωρώ ότι αν είμαστε πολύ στοχευμένοι στις συζητήσεις μας θα είμαστε σε θέση να διαχειριστούμε καλύτερα τον χρόνο μας. Υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι είχαν αποφασίσει να ζητήσουν το λόγο, αλλά ίσως να ζητήσουν το λόγο και άλλοι που βρίσκονται στην αίθουσα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τώρα να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μιχαήλεβα. Θα υπάρχει όριο, για, χρονικό όριο για τις παρεμβάσεις κατά τη διάρκεια των συζητήσεων. Τώρα όμως να δώσω το λόγο σε πρώτη φάση στον κύριο Ντεφά, Γενικό Διευθυντή για την Περιφερειακή και Αστική Πολιτική από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μας παρουσιάσει την κυρία ομιλία της συνεδρίασής μας. Uh, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ τα μέλη της Επιτροπής, το Πρόεδρο Βόσνιακ και τα μέλη της Επιτροπής, ε, της Επιτροπής Κοτέρ ως Γενικός Διευθυντής για Περιφερειακά Θέματα. Είναι τιμή μου που μου δώσατε το λόγο και είναι χαρά μου που ε, βλέπω και, τους, και τις δύο επιτροπές από κοινού εδώ. Ο Επίτροπος Χάν σας έδωσε μια καλή επισκόπηση των μεταρρυθμίσεων τα τελευταία πέντε χρόνια. Επίσης σας ενημέρωσε για την κατάσταση στην εφαρμογή του νέου προγράμματος. Τελείωσε ο Επίτροπος Χάν λέγοντας ότι τώρα έχει φτάσει η στιγμή ε, της πράξης. Και γι' αυτό στη σύντομη παρέμβασή μου θα ήθελα να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας στα της εφαρμογής. Θέματα εφαρμογής τα οποία είναι πράγματι κρίσιμα για την επιτυχία των προγραμμάτων αυτών κατά τη διάρκεια της επόμενης περίοδου. Θα αναφερθώ λοιπόν σε τρία θέματα. Το πρώτο και το έχετε αναφέρει και οι δύο συμπρόεδροι, είναι το πώς η ολοκληρωμένη αυτή ανάπτυξη των περιφερειών και των αστικών περιοχών θα ενισχυθεί. Θα μιλήσω επίσης και για την εκ των προσέρων αιρεσιμότητα και μετά μαζί με, τον, ε, με τις παρεμβάσεις οι οποίες να είναι προσανατολισμένες σε αποτελέσματα να δούμε πώς μπορούμε να μεγιστοποιήσουμε την ωφελημότητα των δράσεών μας. Θα αναφερθώ επίσης και στα θέματα των ε, διοικητικών ε, ικανοτήτων ή δυνοτήτων που απαιτούνται για να εφαρμοστούν σωστά όλα αυτά τα μέσα. Ας μιλήσω τώρα για τα νέα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας με τη νέα νομοθετική ρύθμιση για την εφαρμογή της στρατηγικής σε τοπικό επίπεδο, το CLMD δηλαδή τα προγράμματα αυτά των οποίων ηγούνται οι τοπικές κοινότητες. Είναι κάτι το οποίο ε, μπορεί να λειτουργήσει σε τοπικό επίπεδο αντιμετωπίζοντας οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές ε, υποθέσεις. Τοπικές ομάδες που εμπλέκουν εκπροσώπους όλων των τομέων της τοπικής κοινωνίας και των τοπικών συμφερόντων. Αυτό βασίζεται στην εμπειρία την οποία έχουμε σωρεύσει κατά τη διάρκεια της ε, προηγούμενης δεκαετίας και στα πλαίσια του Urban και του Leader. Μετά από τις προκαταρτικές εξημίσεις στα πλαίσια της νέας προγραμματικής περίοδου, μπορούμε να πούμε ότι 16 χώρες έχουν χρησιμοποιήσει τα προγράμματα αυτά περίπου στα 2 δις 1,4 για το κοινωνικό ταμείο και τα υπόλοιπα για το περιφερειακό. Το 90% των πιστώσεων αυτών χρησιμοποιούνται στις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές. Υπάρχουν επίσης και τα ITI, τα ολοκληρωμένα επενδυτικά προγράμματα. Και εδώ έχουμε νέους πολύ ενδιαφέροντες μηχανισμούς απόδοσης των προγραμμάτων αυτών, που επιτρέπουν τον συνδυασμό πολλαπλών προγραμμάτων και προτεραιοτήτων σε, ε, ένα πλαίσιο πληρωμών. Ε, ασχολούνται με την κάλυψη ενός συγκεκριμένου τομέα ή περιφέρειας και τα ITIs δίνουν τον τρόπο για μια πιο ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των τοπικών αναγκών μετά από τις προκαταρτικές αξιολογήσεις τις οποίες έχουμε προβεί, βλέπουμε ότι 21 κράτη-μέλη μέχρι τώρα, καλύπτοντας περίπου το 90% του ευρωπαϊκού πληθυσμού καλύπτουν τα ITIs και για τις αστικές περιοχές ε, στα πλαίσια του άρθρου 7 του κανονισμού του Περιφερειακού Ταμείου αλλά και για άλλα θέματα. Αυτά για το μέσο, τα μέσα τα, τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας. Τώρα, εκ των προτέρων ερεσιμότητα. Υπάρχουν νέοι μηχανισμοί στα πλαίσια των προγραμμάτων αυτών. Ξέρετε ότι οι νομοθέτες έχουν δημιουργήσει την δυνατότητα δίνουν τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να ελέγχονται ε, οι συνθήκες και οι προϋποθέσεις πριν ξεκινήσει η χρηματοδότηση. Έχουμε τρία είδη εκ των προτέρων αιρεσιμότητα. Το πρώτο είναι διακανονιστικού τύπου, δηλαδή συμβατότητα με τις οδηγίες. Δεύτερον, είναι η διαθεσιμότητα των προγραμμάτων πολιτικών και στρατογικών για τη σωστή εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών. Και τρίτον είναι οι διοικητικέ και θεσμικές δυνατότητες και ικανότητες. Οι προϋποθέσεις αυτές λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Είναι κάτι το οποίο είδαμε κατά τη διάρκεια και όλα της προετοιμασίας αυτών των μέτρων. Είναι μια διαδικασία η οποία όμως δεν είναι εύκολη και πάρα πολλές χώρες ε, πρέπει να προτείνουν προγράμματα δράσης με συγκεκριμένες προθεσμίες, γιατί προς στιγμή δεν εκπληρούν πλήρως τις προϋποθέσεις της εκ των προτέρων αιρεσιμότητας, αλλά θα το κάνουν αυτό με τα προγράμματα δράσης το αργότερο το 2016. Πού είναι οι πιο δύσκολοι τομείς, δύο ειδών είναι οι δύσκολοι τομείς. Πρώτον, πλήρης μεταφορά και εφαρμογή των ευρωπαϊκών ρυθμίσεων και οδηγιών και δεύτερον η ανάγκη δημιουργίας μιας περιφερειακής στρατηγικής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρθηκε πρώτα στη στρατηγική και μετά σε προγράμματα, όχι πρώτα σε προγράμματα και μετά σε στρατηγική. Απαιτείται η ύπαρξη λοιπόν μιας γενικότερης στρατηγικής, ιδιαίτερα σε τομείς όπως ε, οι διοικητικές υποδομές, οι μεταφορές και η εκπαίδευση και η υγεία. Θα πρέπει επίσης να είμαστε βέβαιοι ότι τα προγράμματα αυτά εντάσσονται σωστά στην ευρύτερη μεταρρυθμιστική και οικονομική πολιτική της περιφέρειας και της χώρας. Και γι' αυτό ακριβώς εδώ τίθενται και τα θέματα των ειδικών συστάσεων αναχώρα. Μιλάμε για μια διαδικασία η οποία πηγαίνει καλά. Ένα τρίτο σημείο το οποίο συνδέεται με αυτά τα οποία σας ανέφερα τις συστάσεις αναχώρα και την εξάντε ερεσιμότητα. Ε, Είναι το θέμα των διοικητικών ικανοτήτων. Υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν ε, λάβει συστάσεις συγκεκριμένες για τις χώρες αυτές για να βελτιώσουν τις τους, τη διοικητική τους δυνότητα, τις διοικητικές τους ικανότητες και υπάρχουν και εξάντε αιρεσιμότητες στον τομέα των δημοσίων προμηθειών, των κρατικών βοηθειών, ενισχύσεων και υπάρχουν και δυνατότητες βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας και στον τομέα της ε, απασχόλησης. Εν πάση περιπτώσει βλέπετε ότι έχουμε ένα πλήρες μέτωπο μέσων, εργαλείων έτσι ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες των διοικητικών ικανοτήτων, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικές για τα προγράμματα και την εφαρμογή τους. Η εμπειρία μας μέχρι τώρα είναι σαφής. Υπάρχει ε, υψηλότατο συσχετισμός ανάμεσα στην ποιότητα της διοικητικής διακυβέρνησης και την απορρόφηση ε, των πιστώσεων. Η χαμηλή απορροφητικότητα συνάδει με την χαμηλού επίπεδου διοικητική ικανότητα και διακυβέρνηση. Ε, πέραν αυτού άλλωστε και ε, το ελεγκτικό συνέδριο μας υπενθυμίζει σε τακτική, σε αιτήσια βάση ότι στον τομέα των δημοσίων προμηθειών, στον τομέα των κρατικών επιδοτήσεων και ενισχύσεων ε, εκεί ακριβώς ε, υπάρχουν αδυναμίες σε επίπεδο ε, διαχειριστικών αρχών και είναι υπεύθυνες εμπολείς οι αρχές αυτές για τα υψηλότατα επίπεδα λαθών που έχουμε στον τομέα της συνοχής. Έχει σημασία λοιπόν να αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά συγκεκριμένα. Όταν κοιτάει κανείς τα θέματα της διοικητικής ικανότητας μπορεί να τα αναλύσει κάπως επιμέρους διάρθρωση, συστήματα και μέσα. Και στα τρία αυτά υποεπίπεδα μπορούμε μέσω της τεχνικής βοήθειας να συνδράμουμε. Έχει σημασία λοιπόν οι περιφέρειες και τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν την τεχνική ε, βοήθεια, την τεχνική αρρωγή με κατάλληλο τρόπο έτσι ώστε να ενισχύσουν τις διοικητικές τους διαχειριστικές τους ικανότητες. Αυτό στο παρελθόν γινόταν αλλά όχι με στρατηγικό και οργανωμένο τρόπο. Για τη νέα λοιπόν προγραμματική περίοδο η τεχνική βοήθεια και οι πιστώσεις για την τεχνική βοήθεια θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν με στρατηγικό στόχο την βελτίωση της διοικητικής ικανότητας των διαχειριστικών αρχών. Ε, ε, υπάρχουν λοιπόν συγκεκριμένα θέματα για συγκεκριμένες χώρες και ήδη προγραμμάτων υπάρχουν ε, κάποιες ε, δυσκολίες σε επίπεδο ε, διαχειριστικό που έχουν πολύ μεγάλη σημασία για αυτό μισό όπως το περιβάλλον και πολλές χώρες σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν το 11 λοιπόν και εκεί έχουν εντοπιστεί μερικές φορές κάποιες στρατηγικές οι οποίες δεν είναι τόσο ξεκάθαρες όσο ε, εμείς τουλάχιστον θα επιθυμούσαμε. Συνεπώς, το πρώτο θέμα στα πλαίσια της βελτίωσης της διαχειριστικής ε, ικανότητας είναι η τεχνική βοήθεια την οποία μπορεί να δώσουμε, αλλά δεν σταματά εκεί αυτό. Εμείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθούμε να συνεισφέρουμε ενεργά στην βελτίωση της ποιότητας μέσω της δράσης μας. Στην Γενική Διεύθυνση Περιφέρειας, Περιφερειών μάλλον, δημιουργήσαμε εδώ και δύο περίπου χρόνια μια ειδική μονάδα για την ενίσχυση των διαχειριστικών δυνατοτήτων ε, των ε, περιφερειών και των ε, αστικών περιοχών κτλ. Να σας δώσω ίσως κάποια παραδείγματα. Πρώτον, παρέχουμε καθοδήγηση σε όλου σε όλων των τύπων της δραστηριότητες, σε επίπεδο δηλαδή ελέγχου, σε επίπεδο αδειοδότησης, σε επίπεδο εφαρμογής. Νομίζω ότι υπάρχουν αρκετά παραδείγματα εδώ, ένα από αυτά είναι ο τομέας των δημοσίων προμηθειών. Ε, εμείς με πάρα πολύ τρόπο συστήνουμε τρόπους αποφυγής των συνηθέστερων λαθών στον τομέα των δημοσίων προμηθειών. Αυτό είναι καλό που το υπενθυμίζουμε και μάλιστα κατά τη διάρκεια αυτών των ημερίδων θα σας παρουσιάσουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Έχουμε ξεκινήσει επίσης μια ευρύτερη δράση κατάρτισης η οποία ξεκίνησε τον μήνα Ιούνιο και θα τερματιστεί τον επόμενο Μάρτιο. Σε δύο ε, στόχους, με δύο στόχους, καταρχάς προσανατολισμός των νέων προγραμμάτων και δεύτερον βελτίωση της διαχειρισιμότητάς τους. Με αυτά τα πιλωτικά προγράμματα ε, θα έρθουμε σε επαφή και ελπίζουμε θα βελτιώσουμε 340 τοπικούς διαχειριστές. Ξεκινήσαμε επίσης διασκέψεις και εργαστήρια για την καταπολέμηση της διαφθοράς και των απατών. Εδώ το κάνουμε σε συνεργασία με άλλες γενικές διευθύνσεις μεταξύ των οποίων και της ΟΛΑΦ. Μέχρι τώρα έχουμε οργανώσει έξι συμβάντα, έξι συνεδριάσεις με άνω των 500 συμμετεχόντων και θα ακολουθήσουν και άλλες. Πρόκειται για μια πολύ πρακτική βοήθεια λοιπόν. Υπάρχουν ε, επίσης κοινέ δράσεις και με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Το 2013 τα χαρτοφυλάκια τα οποία στηρίχθηκαν με αυτόν τον τρόπο αφορούσαν πάνω από 600 προγράμματα και έφταναν το ύψος των 60 εκατομμυρίων. Και τέλος, προετοιμάζουμε ένα σύστημα ανταλλαγής απόψεων εθνικών εμπειρογνωμόνων, το λεγόμενο Regio Peer-to-Peer, -peer, μεταξύ ομολόγων δηλαδή, ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα σε διαχειριστικές αρχές, πιστοποιητικές αρχές και ελεγκτικές αρχές. Αυτά θα επιτρέψουν <clears throat> και στις ασθενέστερες διοικητικά τοπικές αρχές να ωφεληθούν από τις εμπειρίες των υπολείπων ίσως πιο αποτελεσματικών. Λοιπόν, προχωράμε και προς την κατεύθυνση αυτή στην παρούσα φάση. Βλέπω ότι δεν έχω πλέον χρόνο. Νομίζω ότι σας έδωσα τις βασικές γραμμές των δραστηριοτήτων μας σε έναν πάρα πολύ βασικό τομέα των της διαχειριστικής ικανότητας. Ολοκληρώνω εδώ και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Thank Σας ευχαριστώ πάρα πολύ θεωρώ ότι αυτό είναι σημάδι καλή συνεργασία ανάμεσα στην Επιτροπή Ρέτζι και ε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν χρειάζεται καν ε, να ε, μιλάμε, καταλαβαίνουμε από τα βλέμματα ακριβώς τι εννοούμε όταν πλησιάζει η ώρα να κλείσουμε. Εν πάση περιπτώσει, έχει έρθει η ώρα τώρα για τη συζήτηση. Παρακαλώ τα μέλη και των δύο επιτροπών να τηρήσουν το χρόνο ομιλίας. Και σας παρακαλώ, δύο λεπτά για τις παρεμβάσεις σας ο καθένας. Ωραία. Πρώτος ομιλητής είναι ο κύριος ε, Μιχαήλ Σνάιτερ, πρόεδρος ε, του, της ομάδας του ΕΛΚ από την Επιτροπή των Περιφερειών. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, ε, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα αναφερθώ σε αυτό που είπα πριν. Με την ε, νέα πολιτική συνοχή νομίζω ότι έχουμε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα μπροστά μας και ένα φιλόδοξο εργαλείο στη διάθεσή μας. Αυτό είναι αποτέλεσμα μιας καλής και φιλικής συνεργασίας ανάμεσα στην Κοτέρ και την Ρέτζη. Εγώ το τελευταίο διάστημα ήμουν πρόεδρος της Κοτέρ και εκτίμησα την συνέργαση αυτή και ήταν μια εμπειρία που ε, θα έχω και για το μέλλον. Δημιουργήσαμε μια ομάδα εργασίας ad hoc που είχε ως καθήκον την παρακολούθηση των τότε νέων κανόνων. Πώς λειτουργούν στην πράξη αυτά που είχαν μόλις τότε. Ταυτόχρονα να κοιτάει στο το μέλλον ε, τι μορφή θα πρέπει να έχουν τα πράγματα μετά το 2014 με βάση τις εμπειρίες ε, που έχουμε συλλέξει. Και έτσι η ομάδα αυτή στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό στις εμπειρίες των περιφερειών. Για την Επιτροπή των Περιφερειών ε, θα ήθελα να προτείνω και στο μέλλον να συνεχίσουμε με τον τρόπο αυτόν την του χρόνου ενδεχομένως να δημιουργήσουμε μία ομάδα η οποία καθήκον θα έχει να παρακολουθεί τους νέους κανόνες. Όλα αυτά που σήμερα ακούγονται τόσο ωραία λειτουργούν στην πράξη. Τι λειτουργεί, τι δεν λειτουργεί, τι εμπειρίες θα έχουμε στην πράξη και να προτείνει στο μέλλον να βελτιώσουμε το τάδε ή το δίνα πράγμα. Πολυπλοκότητα της ε, διοικητικής ε, προσπάθειας, αυτό είναι ένα θέμα με το οποίο σίγουρα θα πρέπει να ασχοληθούμε και δεύτερον ως προς το περιεχόμενο στο μέλλον οι δημογραφικές εξελίξεις τι επιπτώσεις θα έχουν στην πολιτική συνοχή και πώς μπορεί να αντιμετωπίσει αυτή την πρόκληση η πολιτική συνοχή στο μέλλον. Ήθελα να ανακοινώσω τα δύο αυτά θέματα σήμερα και ελπίζω στο μέλλον να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την εντατική συνεργασία που είχαμε και στο παρελθόν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δίνω το λόγο στον κύριο Etheridge. Ευχαριστώ. Καταρχάς ε, θέλω να επενέσω όλους ε, για τα πολύ θετικά αισθήματα που ε, διαπίστωσα ότι υπάρχουν σήμερα. Όλοι έχουν καλές προθέσεις και ήταν πολύ θετικό. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μια, ένα απόφαγμα που λέει ότι ο δρόμος για την κόλαση είναι στρωμένος με καλές προθέσεις. Ελπίζω λοιπόν να μην μείνουμε μόνο σε αυτές. Μιλήσαμε για το τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Ε, ωστόσο, το συζητάμε αυτό ε, στο κέντρο της εξουσίας, σε αυτό το ε, κάστρο των καλών προθέσεων. Συμφωνώ με τον τελευταίο μιλητή ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε... Μάλλον άκουσα αυτά που είπε ο τελευταίος ομιλητής να ενισχύσουμε την διοίκηση, αλλά δεν έχω την εντύπωση ότι αυτό φτάνει στους ανθρώπους σε τοπικό επίπεδο. Εγώ είμαι Ευρωβουλευτής για τα West Midlands της Αγγλίας και ε, εγώ ιδιαίτερα σωστό βρήκα αυτό που άκουσα για τις περιφέρειες και τις αστικές περιοχές. Στη συζήτησή μου γίνεται, υπάρχει μια πολύ εντατική συζήτηση σχετικά με το Birmingham ε, και το εκτεταμένο Birmingham. Ε, μερικοί θεωρούν ότι αυτό είναι καλή ιδέα, αλλά οι άνθρωποι που θα προσχωρήσουν σε αυτήν την μεγάλη περιοχή πώς θα νιώσουν, πόσο μάλλον που η περιοχή αυτή είναι γνωστή ως η μαύρη χώρα ε, λόγω του βιομηχανικού παρελθόντος της. Ε, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πολύ ισχυρή περιφερειακή ταυτότητα. Δεν θέλουν να προσχωρήσουν στο Μπέρμιχαμ, ούτε ε, οι πολίτες του Μπέρμιχαμ θέλουν να ε, τους έχουν μαζί τους. Πολλοί κόσμος λοιπόν δεν θέλει τέτοια πράγματα. Ε, ήθελα λοιπόν ε, να κάνω την παρέμβαση αυτή. Ξέρω ότι δεν μπορώ να σας εμποδίσω να κάνετε αυτά που θέλετε, αλλά ήθελα να σας ενημερώσω ότι υπάρχουν ε, κάποια προβλήματα με τις ιδέες που διατυπώνουμε εδώ πέρα. Πιστέψτε με, υπάρχει κόσμος που τις αντιπαθεί ιδιαίτερα τις ιδέες αυτές. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να δώσω το λόγο στον Σερ Άλμπερτ Μπορτ Ευχαριστώ Μάρικ και θα ήθελα να αναφερθώ στις προτάσεις του Μίχαελ Σνάιντερ σχετικά με τη δημιουργία ε, ενός μόνιμου φορέα ε, των Επιτροπών ε, Ρέτζι και Κοτέρ. Πιστεύω ότι κάτι τέτοιο θα μας οδηγήσει σε καλύτερη κατανόηση της εφαρμογής των προγραμμάτων αυτών και θα επιτρέψει στην Επιτροπή Ρέτζι μαζί με την Επιτροπή να διασφαλίσει τον μελλοντικό προσανατολισμό των εργαλείων για την ε, πολιτική συνοχής. Άκουσα προσεκτικά αυτά που είπε ο Γενικός Διευθυντής για την Περιφερειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα ήταν πολύ χρήσιμο τα κράτη-μέλη που δεν συμμορφώνονται με την εισαγωγή των ITI ε, ε, να αναφερθούν. Ε, μπορώ να σας αναφέρω ένα από τα κράτη αυτά, το Ηνωμένο Βασίλειο. Και αν σκεφτούμε τον πληθυσμό του Ηνωμένου Βασιλείου, τα διαρθρωτικά ταμεία και ταμεία επενδύσεων διανέμονται από φορείς ε, που δεν ε, λογοδοτούν και που δεν είναι ενδιάμεση ε, φορείς, αλλά θα αποτελέσουν παρόλα αυτά την βάση για την κατανομή των πόρων. ITI υπάρχει μόνο στο Cornwall. Και γι' αυτό ο στόχος που είχαμε εδώ και πολλά χρόνια στην Επιτροπή των Περιφερειών να δημιουργήσουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τις εδαφικές δραστηριότητες υποσκάπτεται, υπονομεύεται από ε, την ε, αντίσταση στην προσέγγιση ITI. Ο λόγος που πιστεύω ότι είναι χρήσιμο να υπάρχει μόνιμος φορέας ε, των Επιτροπών Ρέτζι και Κοτέρ είναι ότι έτσι θα μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε την τεχνογνωσία των τοπικών αρχών. Έχουμε την τεχνογνωσία αυτή και μαζί με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα μπορούμε σε ε, ε, μηνιαία ή διμηνιαία βάση να επανεξετάζουμε τα προγράμματα και να βλέπουμε πού βρίσκονται οι ενδεχόμενες αδυναμίες τους. Πιστεύω ότι αυτό θα το επικροτούσε και η Επιτροπή των Περιφερειών και ελπίζω να είναι θετική ανταπόκριση στο αίτημα του Μάικλ και το δικό μου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Ντέλη. Σας ευχαριστώ πρόεδρε, θα μιλήσω ουγγρικά. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ. Θα ήθελα και εγώ να συμφωνήσω με τους ε, προλαλήσαντες. Οι οποίοι και τόνισαν και στην προηγούμενη συνεδρίαση ότι είναι σημαντικό η απορροφητικότητα των περιφερειών και των ε, πόλεων να ενισχυθεί. Ο κύριος Γενικός Διευθυντής της ε, Γενικής Διεύθυνσης Ρέτζη υποστήριξε ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πολύ πρόθυμη και δραστήρια προς την κατεύθυνση αυτή σε ό,τι αφορά τις περιφερειές και τις ε, τοπικές κοινότητες και ότι υποστηρίζονται οι θύνοντες σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό αυτό που δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΩΣΑ. Μίλησε για ένα διαδραστικό φάκελο. Μια βέλτιστη, λοιπόν, μια βάση δεδομένων για τις βέλτιστες πρακτικές σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση των μέσων για την πολιτική συνοχής θα μπορούσαμε να έχουμε μια τέτοια βάση δεδομένων. Θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Να υπάρχει μια επισκόπηση για τις πρακτικές αυτές που υφίστανται, όχι μόνο βάσει των δικτών που χρησιμοποιούνται από το ΩΣΑ, αλλά και από, τις Ευρωπαϊκή, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, προκειμένου να δημιουργηθεί μια εικόνα ενιαία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Χρήσιμο θα ήταν επίσης να αυξήσουμε αυτές τις εμπειρίες σε ό,τι αφορά τις αναδιαρθρώσεις, για παράδειγμα, που γίνονται στα κράτη-μέλη. Συχνά έχουμε προγράμματα τέτοια αναδιάρθρωσης στις περιφέρειες και θα μπορούσαμε λοιπόν στην περίπτωση αυτή να βασιστούμε στις προηγούμενες εμπειρίες των κρατών μελών με μια τέτοια βάση δεδομένων θα μας επέτρεπε να εξετάσουμε ποιες είναι οι ποιοτικές διαφορές μεταξύ των διαφόρων περιφερειών. Γιατί κάποιες περιφέρειες θα πηγαίνουν καλύτερα σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος, και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Βοσνιάκ. Ναι, έχω μια λίστα με νέα ομιλητές. Εννέα άτομα θέλουν να πάρουν το λόγο. Μπας Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή της Επιτροπής των Περιφερειών για την νέα ενοποιημένη ατζέντα για τις πόλεις. Οι πόλεις έχουν αναπτυχθεί και αποτελούν τους οικονομικούς κινητήρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για μια μεγάλη φάση αλλαγών και μια μεγάλη φάση προκλήσεων με νέους πολίτες με τη μετανάστευση, με την ενέργεια των νέων. Η οικονομική καινοτομία λοιπόν και η διαφορετική αντιμετώπιση της ενέργειας είναι πολύ σημαντική πτυχές, γιατί στις πόλεις συμβαίνουν όλα αυτά. Σε 20 χρόνια 85% του πληθυσμού θα μείνουν σε πόλεις. Είναι λοιπόν χρήσιμε οι πόλεις για το πόσο θα είναι καλό ο επόμενο αιώνα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να δώσουμε πιο πολύ λοιπόν προσοχή στην αστική διάσταση και στη αφορά την ευρωπαϊκή πολιτική και τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Και είναι πλέον, έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου να δημιουργηθεί μια λευκή βίπλος, βίβλος για την ευρωπαϊκή ατζέντα. Γι' αυτό λοιπόν ζητώ από τους συναδέλφους στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του Κοινοβουλίου να υποστηρίξουν αυτή την πρωτοβουλία και μία ερώτηση προς την κύριο Ντεβάς. Τι θα γίνει με αυτή τη λευκή βίβλο, μπορούμε να την περιμένουμε επιτέλους. Thank you. Σας ευχαριστώ. Άλλος κανείς από την Επιτροπή Ρέτζι. Όχι. Κύριε Βόσνιακ, γιατί και σας ομιλητές τώρα. Κίμερ. Θέλετε να πάρετε το λόγο. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω τον προηγούμενο μιλητή για τα σχόλιά του. Αλλά θα πρέπει επίσης να δούμε τι γίνεται με τις περιφέρειες που δεν εντάσσονται στις αστικές και περιαστικές περιοχές. Αυτό που έχει αρκετή σημασία είναι να θυμηθούμε αυτά τα οποία είπε και ο κύριος Γκουρία και γενικά το τι λέει για τις περιφερειακές μορφές ανάπτυξης ε, ο ΩΣΑ. Έχουν μία αιμονή με την λεγόμενη πολυδιάσπαση των τοπικών αρχών. Εγώ τον φυσβητώ αυτό. Οι Ηνωμένε Πολιτείες έχουν ένα από τους πιο υψηλούς αριθμούς στον κόσμο τοπικών αρχών διαφόρων μεγεθών σε παγκόσμιο επίπεδο. Και διαρωτώνται σε ποιο βαθμό η διάρθρωση αυτή είναι οικονομικά βιώσιμη. Γι' αυτό λοιπόν η πολυδιάσπαση σαν λέξη δεν είναι σωστή εδώ. Σαν παράδειγμα ε, υπάρχουν ε, λογικές οι οποίες πιστεύουν ότι για να μπορέσει να λειτουργήσει η οικονομία αποτελεσματικά απαιτείται ένα απολύτως συγκεντρωτικό σύστημα όπως και μια δικτατορία ίσως. Δεν μπορεί βέβαια να είναι έτσι τα πράγματα. Συνεπώς λοιπόν δεν πρέπει να υποστηρίζουμε εδώ αντίθετα πράγματα. Ναι μεν λέμε το λιγότερο, το μικρότερο είναι το καλύτερο αλλά παρόλα αυτά θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και να μην κάνουμε προτάσεις που μπορεί να αδυνατίζουν την δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλώς. Κώστα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Tração θα ήθελα να εκφράσω και εγώ την δυσαρέσκειά μου για τις διαφορές που ακούμε εδώ από τους διάφορες εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από τις βασικές αρχές ε, της σωστής περιφερειακής πολιτικής. Διαρωτώ με πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέγραψε μια εταιρική σχέση με την Πορτογαλία στα πλαίσια της οποίας οι τοπικές αρχές δεν έχουν κανένα ρόλο να παίξουν. Καταλαβαίνω όταν μιλάμε για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση ότι προβλέπεται η συμμετοχή των τοπικών αρχών. Όταν όμως προβλέπει ένα μεγάλο πρόγραμμα ανάπτυξης για την περιφέρειά μου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι πόλεις μπορούν να απορροφήσουν μόνο το 10% των ε, χρημάτων τα οποία προορίζονται για τις αστικές περιοχές. Είναι ακατανόητος, είναι πόσο τρόπος με τον οποίο έχει διαμορφώσει και την άποψη για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση τις προτάσεις υποτίθετου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι υπέρ των ολοκληρωμένων περιφερειακών επενδύσεων Αλλά αν υπάρχουν περιοχές οι οποίες δεν την χάνουν ε, ομοιογένειας διοικητικής, τότε θα πρέπει να επιδιωχθούν διαφορετικές ε, μορφές ενίσχυσης και επένδυσης. Ίσως και με τη χρήση της κοινωνίας των πολιτών και των ακαδημαϊκών ε, θεσμών σε κάθε περιοχή. Συνεπώς λοιπόν αυτά τα οποία λέγονται εδώ σχετικά με τις ολοκληρωμένες περιφερειακές επενδύσεις στην ουσία κρύβονται σε απλές κρατικές επενδύσεις χωρίς τοπικές συμφωνίες, χωρίς τη διαβούλευση και τη συμμετοχή των τοπικών αρχών. Δεν είναι αυτή η σωστή περιφερειακή πολιτική. Θα ήθελα να υπογραμμίσω δύο ακόμη θέματα. Πρώτον, πώς είναι δυνατόν να υπάρχει μια πολιτική για τις αστικές περιοχές εφόσον ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του Ταμείου Συνοχής δεν επιτρέπουν τη χρήση ε, των πιστώσεων αυτών για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδυτικότητας των αστικών περιοχών, εκτός από την λεγόμενη λαϊκή κατοικία και δεν επιτρέπουν επίσης να υπάρχει και σωστή χρηματοδότηση προγραμμάτων κινητικότητας στο εσωτερικό των αστικών περιοχών και ταυτόχρονα στα πλαίσια της καταπολέμησης των συνεπειών των κλιματολογικών αλλαγών δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τις πόλεις διότι παράγουν το 70% των αερίων του θερμοκηπίου και η βελτίωση της αποδοτικότητας της ενέργειας της πόλης υποχρεωτικά περιλαμβάνει παρεμβάσεις στην ε, κατοικία και στις μετακινήσεις. Τελειώνω με μία ερώτηση, διαρωτώ με. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τελικά προωθεί καινοτόμες δράσεις στον τομέα των αστικών περιοχών. Αυτές οι δράσεις δεν χρηματοδοτούνται από τους εθνικούς προϋπολογισμούς αλλά άμεσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πότε σκοπεύει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ε, να φέρει περισσότερες τέτοιες προτάσεις. Σας ευχαριστώ να δώσω το λόγο στον κύριο Στροματοριτσί. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι οι σκέψεις οι οποίες ακούγονται, τουλάχιστον ε, όπως το πιστεύω εγώ, πρέπει να συνδεθούν κάπως καλύτερα μεταξύ τους. Το πρώτο θέμα στο οποίο θέλω να σταθώ είναι η ανικανότητα από πλευράς των τοπικών αρχών και των περιφερειών και αναφέρομαι και στις περιοχές από τις οποίες προέρχομαι εγώ, από τον νότο της Ιταλίας και τις νησιωτικές περιοχές, από την αδυναμία λοιπόν να κατανοήσουμε σωστά τις προτεραιότητες ε, και το νόημα της ευρωπαϊκής παρέμβασης και εκεί δημιουργούνται συγχύσεις και δεν πετυχαίνουμε να πετύχουμε και να εκμεταλλευτούμε την διαθεσιμότητα κάποιων πόρων που θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στην καταπολέμηση της παινίας, στις διαφθρωτικές ελλείψεις κτλ. Νομίζω λοιπόν ότι έχει σημασία εδώ να σημειώσουμε ε, και αυτό το οποίο είπε η Γενική Διεύθυνση Ρέγγιο, η οποία νομίζω ότι είναι αρκετά σωστή και πιο κατάλληλη όταν μιλάει για στρατηγικές προτεραιότητες. Ο συνδυασμός μέσων και ε, προγράμματα εφαρμόσιμα σε μεγάλη κλίμακα αστικές περιοχές και περιοχές ε, της υπαίθρου όχι σε επίπεδο συγκέντρωσης ε, ε, της πηγής των χρηματοδοτήσεων, αλλά σε επίπεδο συντονισμού, σε ένα επίπεδο, σε μια διάσταση που να είναι αντίστοιχη με τις προτεραιότητες τις οποίες έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάζονται αλλαγές εδώ και χρειάζεται επίσης ε, και αλλαγή στις νοοτροπίες και αλλαγή στην κατάρτιση. Πρέπει να υποστηρίξουμε την αηφορία στις αστικές περιοχές και ταυτόχρονα είναι απαραίτητο αυτά τα προγράμματα ε, ανάπτυξης των αστικών περιοχών να χρηματοδοτούνται σε επαρκές επίπεδο από την περιφερειακή πολιτική της Ένωσης και έτσι να διευρύνουμε και το πεδίο εφαρμογής τους, κάτι το οποίο είναι το βασικό τους πρόβλημα σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω σχετικά. Κυρία Πρόεδρε, μέλη της Επιτροπής των Περιφερειών, ε, της Επιτροπής Κοτέρε και της Επιτροπής Ρέτζη. Κυρίες και κύριοι, είναι πολύ χρήσιμο που ε, τα μέλη της ε, ομάδας Άλτε στην Επιτροπή Κοτέρε έχουν τη δυνατότητα να, ανταλλάξουν τις απόψεις τους σχετικά, να δώσουν τις απόψεις τους σχετικά με το πώς οι περιφερειακές αρχές μπορούν να εκμεταλλευτούν καλύτερα τα διαρθρωτικά ταμεία και να δημιουργήσουν εταιρικές σχέσεις. η προτινόμενη κατεύθυνση για, τα, την πολιτική συνοχή στο μέλλον ε, στοχεύουν στην ε, δημιουργία θέσεων απασχόλησης ε, και αύξησης και θα πρέπει να ανταποκριθούν σε πραγματικές ανάγκες και να δημιουργήσουν πραγματικές δυνατότητες ανάπτυξης. Αυτό βρίσκουμε ότι είναι θετικό. Θετικό είναι επίσης ότι μέρος των ταμείων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη των πόλεων, αλλά πιστεύουμε ότι είναι πολύ χαμηλό το σχετικό ποσοστό. Τα νέα εργαλεία είναι θετικά και προσβλέπουμε στις ε, νέες δυνατότητες που μας δίνουν αυτές οι μέθοδοι αλλά θα πρέπει να δούμε πώς θα διαμορφωθεί η συνεργασία. Το τοπικό και περιφερειακό επίπεδο είναι πιο κοντά στους πολίτες και παίζουν σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή της ευρωπαϊκής πολιτικής ε, με στόχο την ευρωπαϊκή ολοκληρώση και την ανάπτυξη όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε τοπικό επίπεδο γίνεται η πρακτική εφαρμογή η πολιτική συνοχής θα πρέπει να αποκεντρωθεί και θα πρέπει να γίνει σεβαστή η αρχή των εταιρικών σχέσεων. Θα πρέπει το τοπικό και περιφερειακό επίπεδο να έχει αυξημένες αρμοδιότητες όσον αφορά την εφαρμογή της πολιτικής συνοχής και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ε, λαμβάνουν υπόψη τους στο τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής ε, των πολιτικών, κάτι που επιτρέπουν οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης ε, και βλέπουμε καλά παραδείγματα και στην Αυστρία και στην Τσεχία και στην Πολωνία. Στην Σουηδία έχουμε εργαστεί πάνω στην ανάπτυξη του συστήματος αυτού και προβλέπεται χρηματοδότηση από τέσσερα διαφορετικά ε, ταμεία, ε, τα οποία είμαστε η μόνη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιλέξαμε. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε λοιπόν ε, την περιφερειακή επιρροή. Και μία ιδιαιτερότητα της Σουηδία είναι το ότι εξετάζουμε τη στρατηγική πριν την εφαρμογή των προγραμμάτων, αλλά η Κομισιόν φαίνεται να δυσκολεύεται να καταλάβει ε, αυτόν τον τρόπο εργασίας. Τέλος, θα θέλαμε επίσης να τονίσουμε το θέμα της απλοποίησης των κανόνων και του εστιασμού στα αποτελέσματα. Θα πρέπει να απλοποιηθούν οι κανόνες για να διευκολυνθούν αυτοί που ζητούν χρηματοδότηση. Θα πρέπει να γίνει σχετικό συντονισμό. Θέλουμε μείωση τη γραφειοκρατία. Πιστεύουμε όμω ότι θα χρειαστεί πολύ περισσότερο περισσότερη τεχνική υποστήριξη για κάτι τέτοιο. Επικροτούμε τους νέους ε, δείκτες ε, της Κομισιόν ε, και τα προγράμματα που, βασίζονται, που, έχουν, που, που στοχεύουν στα αποτελέσματα. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ανάπτυξη και πιστεύουμε ότι είναι θετική η ανάπτυξη σχετικών δικτών. δεν ε, θα πρέπει να δημιουργηθούν νέες απαιτήσει ε, και προϋποθέσεις. Θέλουμε όλα τα προγράμματα και οι επενδύσεις να οδηγούν σε αποτελέσματα. Νομίζω ότι όλοι το θέλουμε αυτό. Θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, οδηγήσει σε ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό διότι για να αναπτυχθεί η Ευρώπη θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να βρίσκεται πιο κοντά στους πολίτες της και γι' αυτό πιστεύουμε ότι πρέπει να έχουμε το CLLD, ε, διότι έτσι βελτιώνεται η εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους πολίτες. Ευχαριστώ πολύ. Thank Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Φαψίκ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι, η σημερινή εκδήλωση είναι πάρα πολύ σημαντική και θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω και τον κύριο Ντεβά. Είμαι κάπως απογοητευμένος σε σχέση με αυτά που άκουσα και σε ό,τι αφορά τα χρονικά τους χρονικούς περιορισμούς που έχουμε. Δεν είναι επαρκή τα δύο λεπτά. Πώς μπορούμε να περάσουμε ένα μήνυμα σε δύο λεπτά. Αυτό εισαγωγικά ήθελα να το πω. Επίσης, σε τι αφορά τον κώδικα συμπεριφορά, σε ό,τι αφορά τις εταιρικές σχέσεις, χαίρομαι που τονίζεται αυτή η διάσταση της εταιρικής σχέσης και είμαι βέβαιο ότι αυτό θα ενισχύσει και τη διαφάνεια αλλά και το ρόλο των πολιτών στην Ευρώπη. Καλώς ορίζω επίσης το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σε ό,τι αφορά τις πράξεις κάτι εξουσιοδότηση τις οποίες υποστηρίξατε. Αυτό ενίσχυσε τις περιφέρειες. Έχουμε αποθέσει πολλές ελπίδες στην προσέγγιση Τη εταιρική σχέση. Ελπίζουμε να επιφέρει μια αλλαγή στην ατροπία και ελπίζουμε τελικά να αποφασίζει ο πολίτη για το ποιε είναι οι ανάγκε τους και το τι θέλει να υποστηριχθεί. Επίση, ελπίζουμε να κινηθούμε προς μια διαφορετική μορφή διαβούλευση. Θέλουμε πραγματικά να λάβει σάρκα και οστά η προσέγγιση αυτή και ελπίζουμε να μπορέσει να πείσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα κρατη σε ό,τι αφορά την προσέγγιση τη εταιρική σχέση ότι θα πρέπει να μπει στο επίκεντρο της πολιτικής και της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στον τομέα της πολιτικής συνεργής και ασφαλώς επιθυμούμε λιγότερα φόβητρα και πιο πολλά κίνητρα. Ελπίζουμε λοιπόν αυτό να ληφθεί υπόψη και από τα κρατημέλη. Αλλά ασφαλώ θα πρέπει να υπάρξει διαχείριση των ταμείων αυτών, των κονδυλίων αυτών. Χρειάζεται καλή διοίκηση και δεν θα πρέπει όμως οι τοπικές αρχές να είναι υπεύθυνε μόνο για την εφαρμογή. Δεν είναι δυνατόν να παραμένει αναξιοποιητό το μεγάλο ποσοστό των μέσων και να μην ακολουθούνται δημοκρατικές αρχές σε ό,τι αφορά το πώς θα διατίθενται τα κονδύλια αυτά. Να ενισχυθούν λοιπόν οι πολίτες, οι τοπικές οργανώσεις, προκειμένου να μπορέσουμε να πετύχουμε αποτελέσματα. Εγώ είμαι από μια χώρα που συχνά προβάλλεται ως υπόδειγμα για την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών μέσων από μια μικρομεσαία ευρωπαϊκή πόλη. Και ελπίζω λοιπόν οι ευρωπαϊκές πόλεις να έχουν τις ίδιες δυνατότητες ανάπτυξης όπως και οι περιφέρειες. Τώρα κλείνοντας να πω το εξή. Θα πετύχουμε την ανάπτυξη αν επικεντρωθούμε στους ανθρώπους. Στην Ευρώπη δεν μπορούμε να επιτρέψουμε για απασχόληση να μην λαμβάνετε στα σοβαρά γιατί κυρίως η ανεργία των νέων είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να καταπολεμήσουμε και ιδιαιτέρως θα πρέπει να σκεφτούμε το μέλλον των παιδιών μας και σε αυτό να επενδύσουμε. Το μέλλον αυτό λοιπόν είναι δυσίωνο. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα έχω ακόμα τέσσερις ομιλητές στον κατάλογο των ομιλητών. Και έτσι λοιπόν δεν θα μιλήσω εγώ, δεν θα κάνω τα καταλεκτικά σχόλια που σκοπεύα να κάνω. Μπράντζερ, Καμαλίο, Μπαγιέρ, Μπενάρ, Έστα, θα πάρουν το λόγο. Πιστεύω λοιπόν ότι Όλοι θα πάρουν το λόγο έτσι. Ο κύριος Μπράνζε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ένα μικρό σχόλιο θα ήθελα να κάνω και δύο επιπλέον σχόλια για την κατάσταση στη χώρα μου, την Τσεχία. Μιλάμε για α, τα λεγόμενα διαχειριστικά μέσα των περιφερειακών ταμείων σε τοπικό επίπεδο. Νομίζω ότι δεν μπορεί να καθορίζονται αυτά μόνο από την εθνική κυβέρνηση, ε, το, το κυβερνητικό επίπεδο συγκεντρωτικά. Πρέπει να εμπλέκονται οι τοπικές και περιφερειακές αρχές. Αυτές είναι που θα προετοιμάσουν τα προγράμματα και αυτές είναι που στην ουσία θα ελέγξουν την εφαρμογή των προγραμμάτων. Ε, βέβαια όταν λέω δεν μπορεί να φανταστώ να συμβαίνει κάτι τέτοιο δεν είναι αλήθεια. Θα μπορούσε να γίνει και θα ήταν αρνητικό. Και γι' αυτό λοιπόν όπως και η Κοτέρ συγκεκριμένα υπογραμμίζει την μεγάλη σημασία που έχουν οι εταιρικέ συμφωνίες και η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση δεν μπορούμε να διαφωνήσουμε με αυτό. Όπως είπε όμως ο κύριος Κώστα, δημιουργούνται προβλήματα και υπάρχει χώρος για βελτίωση. Τώρα για τη χώρα μου, την Τσεχία, ε, εμείς θα χρησιμοποιήσουμε 7 ITIs σε αστικές περιοχές. Πρόκειται για οριζόντια προγράμματα, κάτι το οποίο σημαίνει ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πιστώσεις και από τα κεντρικά προγράμματα και από τα λειτουργικά προγράμματα έχουν σαν στόχο το σύνολο των αστικών περιοχών. Όχι μόνο την ίδια την πόλη, αλλά και τις περιεστικές περιοχές. Εγώ είμαι δήμαρχος ενός χωριού κοντά σε δύο μεγάλες πόλεις και τα προγράμματα αυτά είναι πολύ καλύτερα από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 7-13. Και τώρα έχουμε και τα Local Action Groups, τις ομάδες τοπικής δράσης, οι οποίες είχαν σαν στόχο κυρίως το θέμα της ανάπτυξης της υπαίθρου. Νομίζω ότι οι αλλαγές στα διαφορετικά ταμεία έχουν προκαλέσει δύο προβλήματα. Οι ομάδες αυτές έχουν, παρουσιάζουν πάρα πολλές διαφορές μεταξύ τους. Υπάρχουν άνω των 200 στη χώρα μου άλλες καλύπτουν ε, μια πολύ μικρή περιοχή, άλλες καλύπτουν μια ολόκληρη περιφέρεια. Είναι ασύμβατες αυτές οι ομάδες μεταξύ τους, υπάρχουν ε, τρομερές διαφορές μεταξύ τους, κάποιες λειτουργούν καλά και έχουν μια σωστή στρατηγική, άλλες είναι πολύ πρόχειρες και ad hoc. Συνεπώς λοιπόν υπάρχει ένα πρόβλημα με αυτές τις τοπικές ομάδες ο καθορισμός των δραστηριοτήτων και ο ορισμός του ρόλου αυτών των ομάδων είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει σε επίπεδο βέβαια φιλοσοφικό το χρειαζόμαστε αυτό το μέσο όσο δύσκολο και αν είναι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα κάπως πιο συγκεκριμένα να αναφερθώ σε ένα θέμα ε, και να μην παραμείνω ε, στα θεωρητικά. Εγώ δεν ανήκω στις τοπικές και δημοτικές αρχές. Προέρχομαι όμως από μια περιφέρεια 2.800.000 κάτοικοι και από το 1996 έχει πάρει άνω των 200 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό μας επέτρεψε να περάσουμε από το κατώτερο επίπεδο να φτάσουμε σε υψηλό επίπεδο. Είμαστε μια από τις λίγες περιοχές της Ισπανίας στην Ευρώπη που πέρασαν από την σύγκληση σε ιδιαίτερα αναπτυγμένη περιοχή και μέσω των ποσοστών συγχρηματοδότησης και μέσω της συγκέντρωσης της θυματολογικής και τώρα προσπαθούμε να προσαρμοστούμε στο νέο χρηματοπιστωτικό σενάριο. Προσπαθούμε να το κάνουμε με βάση τα δικά μας δίκτυα. Είμαστε ένα παράδειγμα για το ότι λειτουργεί η πολιτική συνοχής και μπορεί να είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Ε, εμείς έχουμε συγκεκριμένο δίκτυο λοιπόν που πέρασε στην αύξηση του ΑΕΠ ποσοστία από 0,8 σε 1,26. Περάσαμε λοιπόν με τα σωστά χρηματοδοτικά μέσα και στον τομέα του περιβάλλοντος. 11,9 του ΦΕΝΤΕΡ για την εξυγίανση των υδάτινων πόρων κάτι το οποίο συνεισφέρει τα μάλλα στο τοπικό μας ΑΕΠ για την καταπολέμηση της ένδυας και των κοινωνικών ανισοτήτων. Το 30% προέρχεται από τα κοινωνικό ταμείο και είμαστε 18 πόντους άνω αυτών που προβλέπει το κοινωνικό ταμείο και ο κανονισμός του. Και έρχομαι εδώ σε αυτά που έλεγε ο κύριος Σνάιντερ για τα δημογραφικά προβλήματα νομίζω ότι πρέπει να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας σε αυτά τα οποία μπορούμε να κάνουμε τώρα με, τον παρόντα προγραμματισμό και να δούμε όμως τι θα κάνουμε και το 2020 σε επίπεδο προγραμματισμού. Απαιτείται σωστός προγραμματισμός, απαιτείται ένα σωστός πολιτισμός της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών. Έτσι θα πετύχουμε τους στόχους και έτσι θα βελτιώσουμε τα αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Περνάς Σολάς. Oui. Άλιστα κύριε Πρόεδρε. Τέσσερις παρατηρήσει. Η πρώτη, τα ITI. Εγώ συμφωνώ με αυτά που είπε ο Αντώνιο Κώστα. Εγώ έχω συντονίσει για τη Γαλλία την προετοιμασία των διαφθορτικών ταμείων. Η περιφέρεια της Λιών 2 ε, εκατομμύρια κάτοικοι. Δυστυχώς πάρα πολύ περίπλοκο να διαχειριστεί κανείς τα προγράμματα. Αυτό είναι δραματικό. Δεύτερη παρατήρηση. Έχουμε καθυστερήσει ιδιαίτερα, άνω του ενός έτους. Προσπάθησα να εξηγήσω στους συμπολίτε μου ότι τα προγράμματα είναι επιλέξιμα την 1η Ιανουαρίου του 2014. Αλλά να συνειδητοποιήσετε ότι οι καθυστερήσεις πλέον είναι πάρα πολύ μεγάλες και πρέπει να πάμε πιο γρήγορα. Τρίτη παρατήρηση. Έχουμε μπροστά μας μια Ευρωπαϊκή Επιτροπή που σε κάποια σημεία συστηματικά έκανε το αντίθετο αυτόν που προβλέπει ο κανονισμός και χρειάστηκε να δώσουμε μάχες ε, και για την κινητικότητα και για τα PIC έτσι ώστε να ακουστεί η φωνή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής Περιφερειών. Είναι ένα σοβαρότατο πρόβλημα και έχω ξοδέψει πάρα πολύ χρόνο πάνω σε αυτό το θέμα και οι συνάδελφοί μου επίσης. Και τέταρτη παρατήρηση, θεωρώ ότι κάποια στιγμή επιτέλους και εδώ θα συμφωνήσουν όλοι να μπορέσουμε να εξηγήσουμε ότι αυτό το οποίο είναι πραγματική επένδυση για το μέλλον είναι η σωστή επένδυση για την Ευρώπη και όχι μια συμπληρωματική δαπάνη που θα πρέπει να υποστεί ε, τις συνέπειες του συμφώνου. Νομίζω ότι δεν πρέπει φυσικά να ξεφύγουμε σε επίπεδο λειτουργικών δαπανών, όπως το έκαναν και οι Αμερικανοί και το κάνουν και σήμερα, όχι η δεξιά και η αριστερά, όλοι μαζί. Αν δεν το πετύχουμε αυτό, ξέρουμε ότι η Ευρώπη χειροτερεύει και θα χειροτερεύσει ακόμα περισσότερο. Σας ευχαριστώ. Κύριε σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σωστό είναι να ασκείτε κριτική για να υπάρξει νέα κίνηση από την κριτική, αλλά σε ό,τι αφορά την έναρξη των ημερίδων αυτών θα πρέπει να κάνουμε και κάποια θετικά σχόλια και να σκεφτούμε τι έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια. Η συνεργασία μεταξύ των, ε, της Επιτροπής των Περιφερειών και της Επιτροπής Ρέτζη του Κοινοβουλίου, η συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Ρέγγιο έχει βελτιωθεί σημαντικά και η διαμόρφωση και η χρήση των ε, κονδυλίων παρουσιάζει στο παρελθόν πολύ μεγαλύτερα ελλείμματα και έχει βελτιωθεί. Έχουμε λοιπόν νέα εργαλεία τα οποία δεν αναφέρθηκαν σήμερα σε ό,τι αφορά την ε, ενταφική συνεργασία η διασυνοριακή συνεργασία, η διαπεριφερειακή συνεργασία το άνοιγμα των περιφερειών και των κρατών σε κράτη που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά είναι τεράστια επιτεύγματα. Η δέσμευση του Επιτρόπου και του Μελλοντικού Επιτρόπου για θέματα γειτονία ε, με κάνει αισιόδοξο σε ό,τι αφορά τα μελλοντικά του καθήκοντα και θεωρώ ότι έχει μεγάλη σημασία σε ό,τι αφορά την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και σε σχέση με τον χάρτη της πολυεπίπεδης διακυβέρνηση. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να ασχοληθείτε τελικά με το θέμα αυτό στη συνεργασία και με τους εμπεριογνώμονε τη Επιτροπή των Περιφερειών. Και χαίρομαι ιδιαίτερω και ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά τη μακροοικονομική στρατηγική και την ανάπτυξή τη, γιατί είναι η τέταρτη μακροοικονομική στρατηγική Και θα πρέπει λοιπόν να ληφθεί ιδιαίτερο υπόψη είναι αυτή η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση εγκάρσια σε όλες τις πολιτικές. Συνολικά θετικά θα πρέπει να αξιολογήσουμε λοιπόν τις εξελίξεις και να δημιουργήσουμε τις ε, ευκαιρίε για μια πιο συχνή ανταλλαγή απόψεων και σκέψεων μέσα ταξί των Επιτροπών Κότερ και Ρέτζι. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Ντεφά Θέλετε να απαντήσετε σε τρία λεπτά. Thanks, uh, mm, There surely, uh, Ναι. Σίγουρα κάποιες παρεμβάσεις ε, δεν απευθύνονται σε μένα, όπως ε, τα περί ε, κοινή ομάδας ανάμεσα στην Κοτέρ και τη Ρέτζη, αλλά θα ήθελα να πω το εξή και ο κύριος Σνάντερ ήταν ο πρώτος που το ανέφερε. Είναι πολύ χρήσιμο και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ Μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ οι εμπειρίες με τα νέα αυτά εργαλεία. Εμείς κάναμε ό,τι θεωρήσαμε δυνατό για να προωθήσουμε τα μέσα αυτά. Έχουμε κάνει τον γενικό προσανατολισμό, έχουμε προσπαθήσει να πείσουμε ανθρώπους, αλλά γνωρίζετε ότι είναι μια εργαλειοθήκη την οποία διαθέτουμε στα κράτη-μέλη και σε αυτά εναπόκειται και στις περιφέρειες να τα χρησιμοποιήσουν. Νομίζω ότι κάναμε ό,τι μπορούμε και κάποια κράτη-μέλη και κάποιες περιφέρειες τα έχουν χρησιμοποιήσει μεγαλύτερη επιτυχία από άλλα. Ε, και αυτό φάνηκε από τη συζήτηση. Πολύ μας ενδιαφέρει λοιπόν ε, να ακούσουμε αντιδράσεις και γνωρίζετε κι εσείς ότι εκπονούνται μελέτες ε, σχετικά με το πώς λειτουργούν αυτά τα νέα χαρακτηριστικά, οι εταιρικέ σχέσεις πώς λειτουργούν και τα εδαφικά μέσα. Επίσης θα με ενδιέφερε να ακούσω τις εμπειρίες σας ε, στους τομείς όπου ε, έχουμε απλοποιήσει τα πράγματα. Η ηλεκτρονική συνοχή, πώς θα λειτουργήσει. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να ακούμε τις αντιδράσεις αυτών που εργάζονται με τα θέματα αυτά στην πράξη. Άλλο θέμα το οποίο θα ήθελα να αναφέρω, επειδή ε, ε, αναφέρθηκε επανειλημμένα στη συζήτηση, είναι η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Είναι σημαντικό να έχουμε μια διαχείριση της γνώσης, διαχείριση των βέλτιστων πρακτικών. Δεν νομίζω ότι μια συνταγή κάνει για όλους, δεν νομίζω ότι υπάρχει θαυματουργή λύση. Μία βάση δεδομένων μπορεί να είναι χρήσιμη σε κάποιες περιοχές, αλλά για παράδειγμα ένα ζωντανό δίκτυο, μια εκδήλωση όπως η Open Days είναι πολύ χρήσιμα πράγματα. Έχουμε και ένα ψηφιακό δίκτυο Αυτά λοιπόν πρέπει να αναπτυχθούν και όπως σας είπα η ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ ε, διοικήσεων των κρατών μελών και περιφερειακών διοικήσεων είναι μια πτυχή την οποία εξετάζουμε. Τελευταία παρατήρηση. Ε, αρκετοί ομιλητές αναφέρθηκαν ε, στο θέμα των πόλεων. Καταρχάς να πω ότι πάνω από το 50% του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης θα αφορά τις πόλεις. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι πόλεις είναι αρμόδιες για αυτά και για να ενισχύσουμε το ρόλο των πόλεων έχετε πιέσει, η Επιτροπή των Περιφερειών και το Κοινοβούλιο, ε, έχετε ασκήσει πίεση για να έχουμε το 5% στο άρθρο 7. Οι πόλεις προσχωρούν στην εφαρμογή των διαρθρωτικών ταμείων. Και όπως είπε ο Επίτροπος, Χαιρόμαστε που η απορρόφηση ξεπερνάει το 5%. Δεν λειτουργεί το σύστημα αυτό σε όλα τα κράτη-μέλη, αυτό είναι αλήθεια. Νομίζω όμως ότι γενικά είναι θετική η εξέλιξη αυτή. Δεύτερον, όσον αφορά τις καινοτόμες ε, αστικές δράσεις. Να σας ενημερώσω ότι θα έχουμε μία πρώτη πρόκληση ε, εκδήλωσης ενδιαφέροντος ε, μέχρι το τέλος της επόμενης χρονιάς ο προπολογισμό ανέρχεται σε περίπου 350 εκατομμύρια. Θα ξεκινήσει το θέμα αυτό του χρόνου. Και τελευταία παρατήρηση και θα κλείσω όσον αφορά την, το θεματολόγιο για τις πόλεις. Είχαμε ανακοίνωση, δημόσια διαβούλευση, η οποία ουσιαστικά έχει ολοκληρωθεί. Ε, κάποιοι συνεισφορείς είπαν ότι χρειάζονται κάποιες μέρες ακόμα. Το επόμενο βήμα θα είναι να αναλύσουμε τις θέσεις των διαφορών φορέων και κατόπιν η νέα Επιτροπή θα αποφασίσει ποια θα είναι τα επόμενα βήματα στο αστικό θεματολόγιο. Κυρία Πρόεδρε, αυτά είχα να πω εντός του τρίλεπτου που μου δώσατε. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Εκτιμούμε την παρέμβασή σας και ότι τηρήσατε το χρόνο σας. Κύριε και έχουμε από τρία λεπτά ο καθένας. E, ευχαριστώ πολύ. Δεν νομίζω ότι θα εξατλώσω το τρίλεπτο. Είναι πολύ δύσκολο να συνοψίσει κανείς όλη τη συζήτηση. Θίξαμε διάφορα θέματα. Πολύ σαφές εδώ είναι όμως ότι μας ανησυχεί ο χρόνος. Έχουμε καθυστερήσεις τις οποίες θα πρέπει να ξεπεράσουμε. Φτάνουμε στο τέλος της περίοδου των δημοσιονομικών προοπτικών και δεν έχουμε και ε, πετύχει πολλά. Δεν θα έχουμε πετύχει πολλά στο τέλος. Θα θέλαμε να ολοκληρώσουμε τις εργασίες πάνω στα έγγραφα. Αυτό είναι σήμερα το καθήκον μας. Υπόθηκε επανειλημμένα ότι πρέπει να σεβαστούμε τον κανόνα της ε, πολλαπλής διακυβέρνησης, ε, της μοιρασμένης διακυβέρνησης ε, και θα πρέπει να λαμβάνουμε η υπόψη της θέσης των εταίρων μας όταν λαμβάνουμε σημαντικές αποφάσεις και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα ήθελα να τονίσω το θέμα των βέλτιστων πρακτικών. Το να προβάλλουμε τα βέλτιστα παραδείγματα. Είναι πάντα αναζητούμε τα καλά μοντέλα που έχουν δημιουργηθεί σε διάφορα μέρη της Ευρώπης. Είναι σημαντικό να γίνεται ανταλλαγή αυτών και θα ήθελα κλείνοντας να σας ευχαριστήσω για τα όσα είπατε. Έχουμε σημειώσει κάποιες σημαντικές θέσεις. Νομίζω ότι η Κομισιόν έχει αποκτήσει μια συνολική εικόνα των θέσεών μας και νομίζω ότι έχουμε πετύχει πολλά σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε που οργανώσατε αυτή τη συνάντηση. Σας ευχαριστώ για την σύντομη σύνοψή σας. Θα ήθελα να συνεχίσω στα βουλγαρικά. Σπάνια έχω την ευκαιρία να χρησιμοποιήσω τη γλώσσα μου. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για τη συμμετοχή σας στη σημερινή συζήτηση. συζητήσαμε μια σειρά προβλημάτων που θα πρέπει να επιλύσουμε. Παρουσιάσαμε διάφορους τομείς στους οποίους θα πρέπει να ε, εργαστούμε περαιτέρω και θα ήθελα να επισημάνω τρία θέματα που κατά τη γνώμη μου ήταν τα κεντρικά της σημερινής συζήτησης. Καταρχάς θα πρέπει να βρισκόμαστε κοντά στους πολίτες. Θα πρέπει να έχουμε κατά νου τι αποτελέσματα θέλουν να δουν οι πολίτες μας. Τα μεμονωμένα προγράμματα θα πρέπει να τα εξετάζουμε προσεκτικά και θα πρέπει να εξετάσουμε πιο προσεκτικά την χρήση των εργαλείων για τη διαμόρφωση της περιφερειακής πολιτικής. Η περιφερειακή πολιτική φέρνει την Ευρωπαϊκή Ένωση πιο κοντά στο πολίτη. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά εξαρτάται από όλους εμάς που εργαζόμαστε στον τομέα αυτόν, ο βαθμός στον οποίο ε, θα φέρουμε κοντά στον πολίτη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλο θέμα είναι η ολοκληρωμένη προσέγγιση. Είναι σημαντικό να ενισχύσουμε το διοικητικό δυναμικό, να ανταλλάσσουμε βέλτιστες πρακτικές και ε, τεχνογνωσία και να οργανώνουμε προγράμματα κατάρτισης. Έτσι οι Ευρωπαίοι πολίτες θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στις κοινέ προσπάθειές μας για μια καλύτερη περιφερειακή πολιτική, δημιουργία καλύτερων συνθήκων ε, ζωής για τους Ευρωπαίους πολίτες. Έχουμε ήδη εμπειρίες στον τομέα της καλής συνεργασίας. Και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για την συμμετοχή σας στην σημερινή συζήτηση. Ευχαριστώ και τους διερμηνείς, λέει η ομιλήτρια, διότι συνέβαλαν στην αλληλοκατανόησή μας. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους διοργανωτές και σας εύχομαι επιτυχία σε όλες τις μελλοντικές προσπάθειές σας και κλείνω την κοινή συνεδρίαση ε, των Επιτροπών για την ε, Εδαφική Συνοχή και τις Περιφέρειες. Ευχαριστώ.